Well, I think we'll have to make a start, otherwise we will begin to be in... Νομίζω θα πρέπει να αρχίσουμε γιατί ο Δάλος θα έχουμε πρόβλημα χρονοδιαγράμματος σε σχέση με εργασίες άλλων. Ε, θα εγκρίνουμε την μερίσια διάταξη πρώτα απ' όλα. Συμφωνείτε, πολύ ωραία εγκρίνεται. Οι ανακοινώσεις της Προέδρου. Ένα λεπτάκι για το χάσα, τα κατάφερα. Σας υπενθυμίζω ότι αύριο το πρωί και το απόγευμα θα διεξαχθεί η συνεδρίαση στην αίθουσα 5Β001. Οπότε να πάρετε τα χαρτιά σας και τους φακέλους σας μαζί. Ουδάλλως μπορεί να απολέσετε κάποια από αυτά. Στη συνέχεια έχουμε την πρόταση οδηγίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων σε θέση με εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Όλοι Σμίτιν ο εισηγητή μα. Όλοι έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε ήδη κάνει την πρώτη σύσκεψη σκιωδών. Νομίζω ότι μέχρι τούδε ήταν παραγωγικές συζητήσεις και ευελπιστώ ότι θα είναι καλή και ικανοποιητική συμφωνία. Το βασικό ζήτημα φυσικά είναι αν θα πρέπει να έχουμε δεσμευτικό στόχο 40% ή όχι. Όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέσσερις εναλλακτικέ λύσεις υπάρχουν. Να καταστήσουμε αυστηρότερο το κείμενο της Επιτροπής, να έχουμε πραγματικές ποσοστώσεις. Δύο, να παραμείνει ως έχει η πρότασή της. Τρίτο, να διατηρήσουμε στου δεσμευτικούς στόχους, αλλά με τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα. Τέταρτον, ε, μία νέα αρχή, ε, συμμόρφωση ή παροχή εξηγήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ε, πρόκειται για την αύξηση προσώπηση ε, των γυναικών ε, σε υψηλόβαθμες θέσεις για να μην εστιάσουμε μόνο σε διοικητικό συμβούλιο. Πολλές εταιρείε προσλαμβάνουν πρώην εκτελεστικούς διευθυντές στο διοικητικό συμβούλιο. Επιθυμούν μεγαλύτερη πρόοδο, αλλά όχι ακολουθώντας την top-down προσέγγιση από τα πάνω προς τα κάτω. Επίσης υπάρχουν μεγάλες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και η πρόταση που κάνω συνεπάγεται θα επιβληθούν δεσμευτικοί στόχοι και θα αναλυθούν δράση από τις εταιρείες σε επίπεδο εκτελεστικών αλλά και μη εκτελεστικών θέσεων, σε επίπεδο διαφάνειας. Οι επενδυτές και οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξακριβώσουν τι συμβαίνει σε περίπτωση της εκπροσώπησης, στον τομέα μάλλον της εκπροσώπησης των δύο φύλων. Πρέπει επίσης να θυμόμαστε, δεν είναι ίδια όλα τα καθεστώτα αυτορύθμισης. Το νορβηγικό παράδειγμα με τις δεσμευτικές ποσοστό ε, δεν είχε την αντίκτυπο που μας ε, είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν διαβάζω την πρόταση του κυρίου Γκίγκολτ βλέπω ότι υποστηρίζουν ε, το θέμα των δεσμευτικών ποσοστώσεων η κυρία Βόρτμαν Κόλλο και ο κύριος Φόξ από τους συντηρητικούς όλοι οι σκιώδεις φαίνεται να ακολουθούν μάλλον το δικό μου προσανατολισμό. Παιδί εφαρμογή. η κυρία Κράτσα θέλει να συμπεριληφθούν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην τροπολογία υπαριθμών 164. Εγώ πιστεύω πιστεύω ότι αυτό είναι μάλλον υπερβολικό και μη, συνεχής μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού άκθους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα η κυρία Ντατή στη δική της τροπολογία 167 θέλει να συμπεριλάβει και ε, τα εκτελεστικά στελέχη ε, το, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε μονομένες δεσμεύσεις. Διάφορες τροπολογίες από άλλους όπως από τον κύριο Λούντβικσον, Γκουλάρε και από τον υποφαινόμενο ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθεώρησε τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν συγγνώμη, και οι μη εισηγμένε εταιρείε. Ε, άρθρο 4, ε, μάλλον το πιο σημαντικό άρθρο, έχει ιδιαίτερη σημασία, υποστηρίζω τι τροπολογίες των κλίν Τρεμόζα, Γένσεν, Τούρβαλς και Φέιου. Πολλοί από εμά υποστηρίζουμε ότι θα πρέπει να δημοσιεύονται οι πληροφορίε από τι εταιρείε για τα μέτρα για την βελτίωση τη ισορρόπηση των δύο φύλων και στι ετήσιε εκθέσει του αλλά και στου ιστοτόπου του. Ο κύριο Γκίγκολ και ο κύριο Λούδιξον, τροπολογίε 201 και 203 ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση. Πολύ σημαντικό το σημείο. Επίση, ο καταναλωτή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγξει το τι πράττουν οι επιχειρήσει, όπω προείπα. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες που ακολουθούν σωστή κατεύθυνση με τη διαγραφή του εδαφείου 4-5 που αντιστρέφει το βάρος απόδειξης για τις εταιρείε για να αποδείξουν την αθωότητά τους εισαγωγικά για την μη έγκριση ενός επιλέξιμου υποψηφίου. Είναι μια καλή πρόταση στους πράσινους, στους φιλελεύθερους, στους και στο ΕΛΚΑ. Πολλοί θέλουν να καταργηθεί η εξαίρεση σε τομείς όπου ε, το εκπροσωπούμενο φύλλο αντιστοιχεί σε λιγότερο από 10% του εργατικού δυναμικού. Νομίζω ότι εύκολα θα το πετύχουμε αυτό. Κυρώσει. Όταν μιλάμε για τι κυρώσει, κατάλαβα ότι πολλοί θέλετε να έχουμε ισχυρότερε ε, ε, κυρώσει. Ε, Βεβαίω υπάρχουν και νομικά κολλήματα, όπω τι τροπολογίε του κ. Γκέκολ 2.28 και 2.30. Κάποιε είναι δυσανάλογα απαιτητικέ, όπω αυτέ του κ. Λούντβινγκσον, του Σουηδού φίλου μα, που προτείνει ε, την πρώτη λύση για τις εταιρείε. Ε, θα κάνουμε βέβαια προσπάθειες ε, ούτως ώστε να θεσπιστούν αρκετά αυστηρές και σκληρές κυρώσεις. Εν κατακλείδη, Πρόεδρε. Ελπίζω και εργάζομαι επ' αυτού. Θα καταλήξουμε σε ευρύτατη συμφωνία, διότι είναι άκρο πολιτικό το ζήτημα. Θέλουμε να διατηρηθεί μια ισόρροπη προσέγγιση και θυμηθείτε ότι ε, είναι μάλλον ε, διαρθρωτικό το θέμα, ούτω ώστε να μετάσχουν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων οι γυναίκε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα, ούτω ώστε να υπάρχει καλύτερη συμφιλίωση οικογενειακή ε, και επαγγελματική ζωή, όχι μόνο με το θέμα τη εκπροσώπηση αντιμετώπιση των δύο φίλων ε, στις επιχειρήσεις αλλά γενικότερα στην κοινωνία και γνωρίζετε ότι ακόμη και στα δικά μας ε, θεσμικά όργανα υπάρχουν δυσκολίες σε σχέση με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ο Ζαν Πολ θα αντικαταστήσει την Κορίν. Έρχεται. Ας περάσουμε στο μεταξύ, στον επόμενο. Όχι, εδώ είναι. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον εισηγητή, το βασικό πρόβλημα αυτής της έκθεσης είναι το άρθρο 4, όπου πρέπει να αποφασίσουμε τι μέτρα θα προωθήσει η ΕΚΟΝ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περαιτέρω συζήτηση ε, στη συνάντηση των σκιωδών που θα έχουμε και αύριο, γιατί μετά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων δεν είμαι σίγουρη ότι συγκλίνουν οι απόψεις μας. Να σας εξηγήσω λίγο την θέση των σοσιαλιστών. Πιστεύουμε ότι το 40% των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια είναι πολύ σημαντικό αν θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο προς την πραγματική ισότητα και τη δημοκρατία. Ο στόχος μας ε, είναι να έχουμε μέτρα που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, μεταξύ των μη εκτελεστικών και εκτελεστικών διευθυντών εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και σε μεταγενέστερη φάση και μεγάλων ε, μη εισηγμένων εταιριών. Πιστεύουμε ότι τα δεσμευτικά μέτρα είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε το στόχο μας και πιστεύω ότι αυτή είναι η βασική διαίρεση που υπάρχει μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Εγώ ε, συντάσσουμε προσωπικά με τον εισηγητή. Ε, τα δεσμευτικά μέτρα είναι και αποτελεσματικά και γρήγορα και μας επιτρέπουν τώρα να πετύχουμε κάποιες αλλαγές. Ενώ τα προαιρετικά μέτρα έχουν όντως αυξήσει, ε, έχουν αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια αλλά όμως ε, η επίπτωσή του είναι βραδύτερη. Το παράδειγμα τη Νορβηγία είναι ένα καλό παράδειγμα επιτυχού εφαρμογή. Έχουμε θεσπίσει εκεί το, την ποσόστοση του 40% το 2006 και τώρα ε, έχει τι περισσότερε γυναίκε η Νορβηγία. Ε, μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να πετύχει το στόχο του 40% η Νορβηγία. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα και εγώ είμαι και μέλο τη επιτροπή Γυναικών εξάλλου και πάντα ακούω αυτές τις στατιστικές για, τις, για την εκπροσώπηση των δύο φύλων και με εντυπωσίασε το παράδειγμα της Νορβηγίας. Πραγματικά η Νορβηγία είναι ένα βήμα προς τα, πιο μπροστά από τους υπόλοιπους ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Έχουν πολλές γυναίκες ε, και από άλλα κράτη-μέλη που είναι επιτυχείς ε, στις είχαν επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στη χώρα τους και μπήκαν σε διοικητικά συμβούλια νορβηγικών εταιριών. Μπορούμε να βρούμε λοιπόν ικανέ γυναίκε με προσόντα για αυτέ τι θέσει, αν τι ψάξουμε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το στόχο του 40%. Ε, δηλαδή θέλουμε ποσόσταση για τι γυναίκε. Από την άλλη, καμία χώρα που έχει χρησιμοποιήσει μόνο τα προαιρετικά μέτρα δεν έχει επιτύχει ούτε καν το στόχο του 30% των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Πόλο δε μάλλον το στόχο του 40% που θέλουμε να πετύχουμε την πρόταση τη Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να τονίσω ότι το χάσμα των δύο φύλων και εκπροσώπησή τους στα διοικητικά συμβούλια είναι θέμα και οικονομικών επιδόσεων και δικαιοσύνης και δημοκρατίας. Γι' αυτό πιστεύουμε στο, στους σοσιαλιστές ότι θα πρέπει να έχουμε διαφανείς διαδικασίες επιλογής με βάση συγκεκριμένα κριτήρια υποστηρίζουμε τις ποσοστώσεις για τα μη εκτελεστικά και εκτελεστικά στελέχη και πιστεύω ότι θα, μας, θα βοηθήσει αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό σε εποχή κρίσης εξάλλου. Για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι εταιρείε, θα πρέπει να αναδιοργανώσουν εντελώ τις πρακτικές τους, τις επιχειρηματικές πρακτικές που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Πιστεύουμε επίσης σε ισχυρότερες κυρώσεις για εταιρείε που δεν σέβονται το στόχο του 40%. Θέλουμε επίσης να α, τις αποκλείουμε από τους δημόσιους διαγωνισμούς και τις κρατικές προμήθειες αυτές τις εταιρείε που παραβιάζουν αυτό το στόχο. Τελευταίο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν πραγματικά αρκετά φιλόδοξη. Αν αποδυναμώσουμε την πρόταση και άλλο της Κομισιόν, που δεν ήταν ούτε καν φιλόδοξη, τι θα, τι θα καταφέρουμε να πετύχουμε τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει πραγματική πρόοδος στην ισότητα με αυτή την στάση. Δεν νομίζω. Ο Ζαν Πολ δεν έχει έρθει, ο Σβέν. Α Σβέν στον κατάλογο. καλά. Τι τυχερό που είμαι, επειδή είναι πολύ περιορισμένο ο χρόνο από ό,τι κατάλαβα από τον εισηγητή, θα ήθελα μόνο να υποστηρίξω τι γενικέ γραμμέ που υιοθέτησαν και οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε και θα ήταν ηρωνικό για μένα εάν το Κοινοβούλιο είχε ασθενέστερη θέση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. σε θέματα περισσότερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το πρόβλημα υφίσταται και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί μόνο με προαιρετικά μέτρα, ούτε με αυτοδεσμεύσεις όσο δεσμευτικές και να είναι αυτές και υποχρεωτικές. Δεν λειτουργεί αυτό όπως προτείνει ο εισηγητής. Και ποιο θα ήταν το επίπεδο, θα ήταν αυθαίρετο. Δηλαδή κάθε εταιρεία θα όριζε, αν ήθελε μόνο 5%, 1% ενδεχομένω. Άλλους τους ικανοποιεί ένα 7%. Ε, δεν ξέρω τώρα, αυτό δεν λειτουργεί. Στη Γερμανία ακριβώς αυτή την εμπειρία είχαμε που αποδείχθηκε και ατελέσφορη. Και τουλάχιστον στη Γερμανία πάνω από 70% του κόσμου έχει βαρεθεί αυτά τα μέτρα που δεν είναι ούτε δεσμευτικά ούτε αποτελεσματικά. Ωστόσο υπάρχει αξία σε αυτή την ιδέα ε, να αποφασίζουν οι εταιρείε ποια μέτρα θα λάβουν για να φτάσουν οι γυναίκες σε περισσότερες ευκαιρίες ε, προαγωγής και ανέλυξης στην ιεραρχία της εταιρεία. Γι' αυτό στις συνεδρίες των σχεδόν εισηγητών έκανα μια πρόταση εγώ. Να παραμείνουμε βασικά στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δεσμευτικούς κανόνες για μεγάλες εταιρείε, αλλά αυτό το πιο προαιρετικό θελούσιο σχήμα να παραμείνει για τις πιο μικρές εταιρείε. Εκεί λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα χωρίς να ε, τους επιβαρύνουμε ιδιαίτερα με κανόνες που μπορεί να μην είναι αναλογικοί για τις μικρές εταιρείες. Οπότε, η ιδέα του εισηγητή νομίζω θα μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να εξυπηρετήσει και να αποτελέσει τη βάση για ένα ευρύτερο συμβιβασμό. Από τη δική μου σκοπιά όμως, και φάνηκε και αυτό από τη σοσιαλίστρια συνάδελφο, ο συμβιβασμός δεν πρόκειται να ευδοκιμήσει ε, βάσει απολύτως προερωτικών και καθόλου δεσμευτικών μέτρων ανεξαρτήτως επίπεδου και ποσοστού και μεγάλες εταιρείες. Okay. Uh, uh, thank you, Chairman. And can I... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε με την νομοδότησή του. Καταλαβαίνω ότι έκανε πολλή προσπάθεια, ούτω ώστε να γίνει αποδεκτό αυτό το νομοθέτημα. Και θα το πετύχουμε και μέσω των συμβαστικών τροπολογιών. Βεβαίω, ακόμα έχουμε τι διαφορέ μα σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι όλοι μα ε, στην Επιτροπή αυτή έχουμε τον ίδιο στόχο. Ο στόχο είναι να αυξήσουμε την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Όλοι θέλουμε ε, δίκαιη και ισότιμη ίση κοινωνία και φυσικά και οι μέτοχοι θέλουν ένα διοικητικό συμβούλιο ποικιλόμορφο που να παίρνει ισορροπημένε αποφάσει. Όπω είπε και η σοσιαλίστρια ε, Ευρωβουλευτή, αν υπάρχει αυτή η ισορροπία στο διοικητικό συμβούλιο, προωθούνται οι καλέ οικονομικέ επιδόσει και είναι προ το συμφέρον τη εταιρεία. Όμω εδώ αρχίζουν ε, να αποκλείουν οι απόψει μα. Γιατί τελικά η εταιρεία είναι στην κατοχή και ιδιοκτησία των μετόχων. Και τελικά απόκειται στου μετόχου να αποφασίσουν πώ οι εταιρείε του την χάνουν διαχείριση. Και είναι αντίθετο κάθετα στη χρήση των νομοθετικών νομοθετικών μέτρων σε αυτόν τον τομέα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε στόχους, όχι ποσοστώσεις, και θα πρέπει να επιτρέψουμε τη φυσική εξέλιξη και αλλαγή των διοικητικών συμβουλίων. Η ισότητα επίσης είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι με τα δεσμευτικά μέτρα δίνουμε μόνο ε, επιφανειακή απάντηση στο πρόβλημα της ισότητας. Πιστεύουμε ότι δεν είναι σωστό να έχουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα, που... γιατί έχουμε να κάνουμε διαφορετικές ε, αγορές εργασίας, τελείως διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον και τελείως διαφορετική δομή και διάρθρωση στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών στις διάφορες χώρες μέλη χώρες μέλη. Επομένως θα πρέπει τα επιμέρους κράτη-μέλη να πάρουν την απαραίτητη δράση που θεωρούν σκόπιμη για τη χώρα του. Σε αυτή τη στιγμή τα διάφορα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα με διαφορετικού τρόπου. Φερρυπίν, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στο Βέλγιο και στην Ιταλία έχουμε νομοθετικά επιβαλλόμενες ποσοστώσεις. Στον Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία και Σουηδία έχουμε αποτελεσματικά μη νομοθετικά μέσα. Ο Σβέν είπε ότι τα προαιρετικά αυτά, οι εθελοντικά μέτρα δεν λειτουργούν. Όχι, λάθος έχει Σβέν. Λειτουργούν λειτουργούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο αριθμός των γυναικών ε, σε εταιρείε που είναι στο φούτσι 100 ε, ε, ανέβηκε από το 12% στο 17%. Μπορώ να τελειώσει παρακαλώ. Α, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Σβέν. Επίσης, με βάση μια έκθεση, φαίνεται ότι θα πετύχουμε ε, στα, μέχρι το 2015 25% των γυναικών και μέχρι το 2020 33% των, των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια εταιριών που είναι εισηγμένες και ε, βρίσκονται στο δίκτυ Φούτσι 100. Αν η γερμανική κυβέρνηση αποφασίσει ότι ας πούμε αυτή η προσέγγιση δεν είναι σωστή για τις γερμανικές εταιρείες, Εσεί στη Γερμανία μπορείτε, α πούμε, αν θέλετε, να προωθήσετε νομοθετική δράση. δεν καταλαβαίνω όμω, γιατί όταν έχουμε μία ε, εταιρεία, μία χώρα όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, που έχει βρει μία αποτελεσματική μέθοδο για να βελτιώσει την κατάστασή τη, γιατί θεωρείτε ότι είναι δηλαδή ε, κατάλληλο να επιβάλλουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα ήθελα να σχολιάσω ε, σύντομα μία τροπολογία την 256 που έχω υποβάλει και που δεν συμπεριλαμβάνεται στους, στις συμβαστικές τροπολογίες. Αυτή η νομοθεσία δεν θα εφαρμοστεί μέχρι η Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, ε, να φτάσει στο πρότυπο, στα πρότυπα που θέλουμε. Στη συνάντηση των σκιωδών, ένας μέλος της γραμματείας είπε ότι δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Για να το πετύχουμε θα πρέπει να αλλάξουμε το καταστατικό Φανταστείτε, ότι δράμα, α πούμε. Είναι τόσο δηλαδή ιερό και απαραβίαστο που δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το περίφημο καταστατικό. Και όμως θέλουμε να νομοθετήσουμε για να αλλάξουμε τη δουλειά και τον τρόπο που λειτουργούν οι ευρωπαϊκές εταιρείε. Τελικά όλα είναι θέμα πολιτικής. Και τελικά η εκλογικά μανιφέστο τη κυρία Ρέντινγκ ε, και όχι τόσο ουσιαστική αλλαγή ε, του αριθμού των γυναικών και μάλιστα εκ των άνω ας καθαρίσουμε λιγάκι τα του οίκου μας πριν αρχίσουμε να επιβάλλουμε νομοθεσία στους άλλους. Ξέρετε, Πρόεδρε, τις απόψεις μου σε αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τον εισηγητή και ελπίζω να πετύχουμε καλό συμβασμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Ζων Πολ μόλις κατέφθασε. Ας μιλήσει για να εκπροσωπήσει την Κορίν. Εν συνεχεία η Άστριντ. Voilà, ça y est. Euh, je ne savais pas que... Δεν ήξερα ότι θα μιλάω εξ ονόματο τη Κορίν σήμερα. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω πιστά το μήνυμα που ήθελα να σα περάσει. Νομίζω είναι, έχει κολλήσει μέσα σε ένα μποτιλιάρισμα και ενδέχεται να μην ε, καταφέρει να καταφτάσει εγκαίρω. Λοιπόν, έξω ονόματο τη Κορίνη, ευχαριστώ τον Όλε Σμιτ για το σχέδιο έκθεσή του. Είναι μια, ένα καλό εφαλτήριο για τι μελλοντικέ συζητήσει μα. Θα είναι πραγματική πρόκληση, λέει η Κορίν, για να καταφέρουμε να έχουμε ευρία πλειοψηφία για την έγκριση της έκθεσης. Ο Όλε όμως έχει, είναι τυχερός, διότι του έχει απόλυτη εμπιστοσύνη η Κορίν. Δύο παρατηρήσεις. Πρώτον για το πεδίο εφαρμογής. Εμείς ε, θέλουμε να διατηρηθεί η εξαίρεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διότι μπορεί να φανεί αυτό για, για, κυρίως για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, να συμμορφωθούν με όλες αυτές τις απαιτήσεις του νομοθετήματος. Ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ως προς τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής για τα διευθυντικά εκτελεστικά στελέχη και το ίδιο ισχύει και για τις εισηγμένες εταιρείε. Στη συνέχεια υπάρχει μια τελευταία πρόταση στο Σμιτ για τις ποσοστώσεις. Ε, πιστεύουμε ότι αποτελεί αυτό καλό έρισμα για τις μελλοντικές συζητήσεις για να καταλήξουμε σε συμφωνία ως προς την εφαρμογή των κανόνων στα ίδια τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Ε, η Κορίν δεν κρίνει απαραίτητο ε, να έχουμε μια γενική προσέγγιση, ούτε χρειάζεται να έχουμε μια ρητή μνήμα στα θεσμικά όργανα τούτου λεχθέντος θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή βάση της οποίας θα πρέπει πρώτα να εφαρμόσουμε εμείς αυτό που κηρύττουμε στους άλλους. Ε, ευελπιστώ ότι δεν εφάν πιστός ως προς το μήνυμα που θέλω να περάσει η Κορίν και το μετέδωσα αποτελεσματικά. Ευχαριστώ η Αστρίντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ θέλω να δώσω συλληπιτήρια στον ε, Όλε Σμιτ ε, ε, γιατί έχει 156 τροπολογίες, είναι 50 δικές το έχει φτάσει στις 206. Αυτές οι τροπολογίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα και σίγουρα θα του δυσκολέψουν τη ζωή. Εγώ ίδια δεν κατέθεσα τροπολογίες για το θέμα διότι γίνεται μια συζήτηση για τη νομική βάση σε εσωτερικές συσκέψεις της ομάδα μας. Αποφασίσαμε να περιμένουμε ε, μέχρι ότου διευκρινιστούν κάποια ζητήματα ω προ τη νομική βάση, διότι... Ε, μιλάμε για τις ε, οδηγίες για δεσμευτικές ποσοστώσεις ε, και είναι λίγο ε, ε, η προσέγγιση αμφισβητείται από κάποιους τέλος πάντων δεν έχουμε καταλήξει σε συμφωνία εγώ ήθελα να σας πω ότι έχω ενδιασμούς ως προς την νομική βάση δεν είμαστε στη Σοβιετική Ένωση είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς να το πω, πώς να το θέσω έχω Έχω αμφιβολίες, αμφιβολίες. Αν είναι σκόπιμο σε μια οικονομία της αγοράς, γιατί εγώ είμαι ο παδός της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, αν λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια θα μπορούσαμε να πούμε στις ε, ε, ιδιωτικές ε, εταιρείες με ποιο τρόπο θα αποφασίζουν τη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων. Είναι μια θέση αρχής αυτή και αναρωτιέμαι αν υπάρχει νομική βάση καν για να παρέμβουμε σε τέτοιο επίπεδο. Επίσης συμφωνώ ότι πρέπει να αρχίσουμε από, τις, από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι οδηγία εδώ, το τονίζω. Θέλω να υπενθυμίσω όμως ε, και απευθύνομαι σε αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει να αρχίσουμε με θελοντικές δράσεις. Σας υπενθυμίζω ότι το 1976, 1976 θεσπίστηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την σύρροπη μεταχείριση ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση της προαγωγής και το καθεξής και επί τη βάση αυτής της οδηγίας που αναφέρω ε, τροποποιήσαμε σύν το χρόνο τις προτάσεις μας. Ε, κανείς δεν ήταν υπέρ των ποσοστώσεων. Εγώ τη δεκαετία του 80 είχα εφαρμόσει στη χώρα μου θετικές δράσεις, ούτως ώστε να προαχθούν ε, ε, όπως πρέπει στις τράπεζες, παραδείγματος χάρη οι γυναίκες. Μετά το 1976 τι έγινε, κανείς δεν έκανε τίποτα. Εγώ το έκανα μέσα σε μια ε, τράπεζα που έφερε την επωνυμία Ευρωπαϊκή Πίστη. Ε, και τότε δεν, ε, στις υψηλόβαθμες ε, στε, θέσεις τελεχών δεν υπήρχαν οι γυναίκες γιατί ποτέ δεν είχε προσληφθεί γυναίκα με πανεπιστημιακό πτυχίο. Έπρεπε να αρχίσουμε πολύ χαμηλά και Όλες Όλε Σμιτ δίκιο έχει. Από κάτω πρέπει να αρχίσουμε και από πάνω. Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των ποσοστώσεων στα διοικητικά συμβούλια στις εισηγμένε εταιρείε. Στο Λουξεμβούργο έχουμε 5-6 τέτοιες. Οπότε τι, θα έχουμε θέσεις ε, ε, για 20-30 γυναίκες. Ε, υπάρχουν πολύ περισσότερες γυναίκες ακόμη και σε τόσο μικρή χώρα που θα άξιζαν μια πιο υψηλόβαθμη θέση. Ε, αν ακολουθήσουμε το νορβηγικό ε, παράδειγμα που το αναφέρουμε επανειλημμένα, στην Ολομέλεια και αλλού έχω τονίσει και εγώ επανειλημμένα ότι έγινε ανάλυση, έγινε έκθεση, μελέτη από μια νορβηγική επιχείρηση ή μάλλον από ένα πολύ σοβαρό επιστημονικό ίδρυμα. Ξέρετε τι διαπίστωσαν. Πριν αρχίσει ο νόμος, ε, υπήρχαν 600 τόσες εισηγμένε εταιρείε. Τρία χρόνια μετά με την εφαρμογή του νόμου κτλ. Εμέναν οι μισέ 300 και κάτι. Όντως είχαμε γυναίκες 300 στο αριθμό στα διοικητικά όχι, 300 θέσει, όχι γυναίκε 300 θέσει. Ε, ε, και ε, είχαμε 70 γυναίκες ε, σε, αυτό το πουλ, σε αυτή την ομάδα θέσεων. λοιπόν, σας είπα ότι εγώ στο Λουξεμβούργο με αυτή την παλιά οδηγία κατάφερα να έχω 20-30 θέσεις. Νομίζω δεν ακολουθούμε σωστό δρόμο. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε τις φυσιολογικές γυναίκες, γυναίκες ε, που συναντούμε καθημερινά ε, και όχι αυτές που κατέχουν τις υψηλόβαθμες θέσεις. Έχουμε πάνω από 250 εκατομμύρια γυναίκες στην Ένωση. Τι μας νοιάζει θα γίνει με τις λίγες χιλιάδες που είναι πάνω πάνω πάνω στην ιεραρχία. Εκείνες που είναι εκεί ξέρουν ήδη τι πρέπει να κάνουν και ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν για να μπουν στα διοικητικά συμβούλια. Εγώ είμαι υπέρ των θετικών δράσεων. Αυτό είναι το σωστό εργαλείο. Και ξέρετε ότι ήδη διώχνουμε τις βιομηχανίες από την Ευρώπη. Και διαβάζω λοιπόν μια τροπολογία και αναρωτιέμαι θα, γιατί θα μείνουν εδώ ε, οι επιχειρήσεις. Τι θέλουν οι πράσινοι πέρα από τις ποσοστώσεις να έχουμε μια πραγματική πολιτική ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών σε όλα τα κλιμάκια της κοινωνίας με καταρτήσεις, με προγράμματα καθοδήγησης για την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, μεγαλύτερη ευελιξία στα ωραία εργασίας, ευέλικτες διατάξεις για τη γονική άδεια. Εντάξει, τα βάλαν όλα μέσα στο ίδιο τσουβάλι. Πολύ ωραία. Εγώ δεν νομίζω ότι εξυπηρετούμε τη θέση των γυναικών με μια τέτοια έκθεση και σίγουρα δεν είναι καλό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν ε, πρόκειται να τα καταφέρουμε με τέτοιου είδους διαβήματα. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει να μιλήσει πριν να επανέλθω στον εισηγητή. Όχι. Όλε Σμιτ. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Όλοι ακούμε ότι θα είναι περίπλοκο αυτό το πράγμα και καταλαβαίνουμε. Αλλά όπως έλεγε και η μητέρα μου, και ποιος σας είπε ότι η ζωή είναι εύκολη. Λοιπόν, αύριο έχουμε την επόμενη μας συνεδρίαση. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς. Τουλάχιστον να βρεθεί κάποια στοιχειώδης πλειοψηφία. Αλλιώς θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για την ψηφοφορία. Δεν έχω άλλα σχόλια πιστεύω. Σας ευχαριστώ για τις ιδέες σας. Α, για την κυρία Λούλινγκ έχω να πω το εξή. Εγώ νόμιζα ότι η επίτροπο από το Λουξεμβούργο είναι από τη δική σα πολιτική οικογένεια. Ναι, αλλά ξέρετε είναι τεράστια η παράταξη μας, λέει η κυρία Λούλη. Εντάξει, το ίδιο ισχύει και για τους φιλελευθέρου. Καλά, δεν είμαστε εμεί τόσο τεράστιοι, αλλά διαφέρουμε ε, στις απόψει, Η πρόεδρος. Μάλιστα. Και έχουμε και πολλά πλοκάμια γενικώ. Ελπίζουμε στις 9 Ιουλίου να είμαστε σε θέση να ψηφίσουμε στην Επιτροπή, στην Καθήλυνα Αρμόδια που είναι η νομική και η γυναικών περίπου στις 14 Οκτωβρίου. Έχετε χρόνο να επιζητήσετε αυτούς τους συμβιβασμούς που χρειάζονται. Αυτά. Λοιπόν, μέχρι τις 4.30 παρακαλώ είμαστε ελεύθεροι. Γιατί ε, έχουμε την κοινή ακρόαση με την άλλη Επιτροπή. Ε, να είστε στην ώρα σας παρακαλώ γιατί όλοι είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις, όλοι θα θέλουν να μιλήσουν για αυτό το θέμα του φίλου, πιστεύαμε. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και ραντεβού στις 4.30.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 think we start uh, Να ξεκινήσουμε γιατί αλλιώς ε, θα έχουμε πρόβλημα χρόνου, ειδικά στο τέλος της συνεδρίασης. Ελπίζουμε και ο Επίτροπος Άντορ τελικά να φτάσει εγκαίρος, ούτως ώστε να εκφωνήσει και αυτό τον λόγο του, μετά τον Όλη Ρεν όμως. Καλωσορίζω τον Όλη στην Επιτροπή μας και Προκαταβολικά καλωσορίζω και τον Επίτροπο Αντόρ. Είναι μια συνάντηση για τις συστάσεις αναχώρα. Είναι η τρίτη δέσμη ετήσιων συστάσεων προς τις χώρες μέλη και στην Ευρωζώνη συνολικά από τη στιγμή που εισήχθηκε το 2010 το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Είναι η δεύτερη φορά που τα σχέδια συστάσεων χώρα λαμβάνουν υπόψη την ε, ενδελεχή αναθεώρηση που έγινε στα πλαίσια της διαδικασίας ε, μακροοικονομικών ανισορροπιών. Και είναι η πρώτη φορά που οι νέες διατάξεις που εισήχθησαν από το 2ΠΑΚ θα εφαρμοστούν. Φερρυπίν, η εποπτεία των ε, ετήσιων σχεδίων προϋπολογισμού, περισσότερες προϋποθέσεις και υποχρέωση προγραμμάτων οικονομικής εταιρικής σχέσης για τα κράτη-μέλη που υπόκεινται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Το Κοινοβούλιο θα δώσει τις απόψεις του για την εφαρμογή του κύκλου του εξαμήνου του 2013 σε μια διαδικασία που ξεκινάει από τώρα και, και η συγγήτρια είναι η Ελίσσα Φερέιρο. Ε, η έκθεσή της θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο. Η Επιτροπή ΕΚΟΝ καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, δουλεύει ε, για τις ε, μελλοντικές μεταρρυθμίσεις ε, της ΟΝΕ και το πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το δημοκρατικό έλλειμμα που, λαμβα... που υπάρχει ε, στα πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πώς θα μπορούσε να πληρωθεί από μια αύξηση των διαδικασιών α, συναπόφασης στα πλαίσια της διαδικασίας του εξαμήνου. Η Κομισιόν επίσης ε, προτείνει ένα κώδικα ε, σύγκλησης, ένα μηχανισμό για κινήτρων για τις μεγάλες εθνικές μεταρρυθμίσεις που θα συμπληρώσει το, την προσπάθεια συντονισμού των οικονομικών ε, πολιτικών ε, με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή και την αποδοχή από τους πολίτες των ε, διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων. Φυσικά το Κοινοβούλιο έχει εκφράσει τις απόψεις του σε κάποιες από αυτές στις συζητήσεις που είχαμε την περασμένη εβδομάδα και κυρίως εξέφρασε τις ανησυχίες του για το κατά πόσο εφαρμόζονται σωστά τα όσα επιβάλλει η νομοθεσία. Πρέπει πρώτα να εφαρμόσουμε σωστά αυτά που λέει η νομοθεσία πριν περάσουμε σε νέο νομοθετικό πακέτο ή προσπάθεια. Τώρα, θα δώσω τον λόγο στον Όλυ Ρεν για 10 λεπτά για να παρουσιάσει τις ε, ειδικέ συστάσεις αναχώρα και συνεχεία θα ακούσουμε τον Επίτροπο Αντόρ όταν τελειώσει όλοι. Όλοι, έχεις τον λόγο. Thanks, uh, thanks, Ευχαριστώ Σάρα, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής των Επιτροπών, καλό σας απόγευμα. Με χαρά βρίσκομαι ενώπιόν σας και σύντομα θα έρθει και ο συνάδελφος Λάσλο Άντερ για να σας παρουσιάσουμε τις ειδικές συστάσεις αναχώρα που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Μαΐου. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού Οικονομικής Πολιτικής ε, διέρχεται τώρα τον τρίτο κύκλο του. Ο σημερινός οικονομικός διάλογος αποτελεί μια ευκαιρία να υπογραμμίσουμε την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το σημερινό οικονομικό πλαίσιο είναι δύσκολο και είναι σαφές ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ξεπεράσουμε την κρίση της ανεργίας και να επιστρέψουμε στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Γι' αυτό εργαζόμαστε για δύο στόχους παράλληλα. Βιώσιμη ε, ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας και σταδιακή εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών. Είναι διτός αυτός ο στόχος και ε, υπόκειται ε, στις φετινές συστάσεις. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι αυτή τη στιγμή εγκριθούν οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα, ε, θα είναι πλέον οι συστάσεις του Συμβουλίου. Άρα δεσμεύονται τα κράτη-μέλη και με συλλογική ευθύνη αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν αυτές τις συστάσεις. Για τρίτη συνεχή χρονιά κάνουμε ειδικέ συστάσεις για την Ευρωζώνη και ε, αφορούν αυτές ζητήματα ε, ιδιαίτερα συνδεδεμένα με το ε, ευρώ όπου έχει την ευθύνη το Eurogroup. Συνδέονται ιδιαίτερα με την ανάγκη σεισμού και πανισορρόπησης της οικονομίας της Ευρωζώνης που ακολουθείται αυτό τον καιρό αφού έχουν συσσωρευτεί μεγάλες και μη ε, βιώσιμες ε, ανισορροπίες στην οικονομία την περασμένη δεκαετία. Αυτή η επανεξορρόπηση λοιπόν και η μεταρρύθμιση είναι σημαντικό να ακολουθείται αποφασιστικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Και εκείνα που έχουν ελλείμματα ε, στις τρέχουσες συναλλαγές τους, αλλά και εκείνα που έχουν πλεονάσματα. Για παράδειγμα, οι στάσεις μας προς τη Γερμανία συμπεριλαμβάνουν ε, βιώσιμη αύξηση των μισθών για να υποστηριχθεί η ε, εσωτερική ζήτηση. Αυτό μεταξύ άλλων απαιτεί μείωση των υψηλών τελών και ε, συνεισφορών των κοινωνικών ασφαλίσεων, ιδιαίτερα για χαμηλόμισθους στη Γερμανία. Παραμένει λοιπόν στόχος μας η εξηγένση των προπολογισμών και οι διορθωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη ε, ακριβώ επειδή είναι πάρα πολύ ψηλό το δημόσιο αλλά και το ιδιωτικό χρέο. Με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταρρυθμίσαμε και μετασχηματίσαμε και το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη ε, για να υπάρξουν οι απαραίτητες προσαρμογές στη διαδικασία εξυγίανσης όταν υπάρξει και αρκετή αξιοπιστία. Ε, έχουν ληφθεί μέτρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχει επιβραδυνθεί ο ρυθμός εξυγίασης. Σύμφωνα ε, με ε, το σύμφωνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στην Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία να εξέλθουν από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ως αποτέλεσμα, ε, μετά τον παρόντα γύρο θα είναι 16 τα κράτη-μέλη και όχι 24 όπως ήταν το 2011. Από 24 σε 16 κράτη λοιπόν στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος μέσα σε μία διετία. Στην οικονομική ανάλυση μας για το Βέλγιο, τις κάτω χώρες και την Πορτογαλία ε, προτείναμε επιμήκυνση της ε, διαδικασίας διόρθωσης για ένα χρόνο και για την Γαλλία Πολωνία, Σλοβενία και Ισπανία για δύο χρόνια. Στο παρόν ευρωπαϊκό εξάμεινο συνδέσαμε ιδιαίτερα και συστάσεις για διορθωτικές ε, αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με αποφάσεις για την εξηγήση του προπολογισμού. Τα κράτη που έχουν λάβει επιμήκυνση μπορούν και θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την ανάσα που τους δίνεται για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους και να ενισχυθούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέψτε μου τώρα να μπω επιμέρους ε, σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη που είναι και επίκαιρα σε σχέση με αυτό, η Ιταλία. Έχει κάνει μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή διαρθρωτική την τελευταία διετία και θα εξασφαλίσει το έλλειμμά της κάτω του 3% ε, επιζητώντας ένα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις είναι κλειδί για την ανάκαμψη στην Ιταλία ε, για να μπορέσει να αποπληρώσει το ε, εμπορικό της ε, χρέος όπως έχει συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε στην οικονομία να επέλθει ρευστότητα και ανάκαμψη. Για τη Γαλλία προτείναμε ε, δίαιτη επιμήκυνση μέχρι το 2015 αντί το 2013. Οι δημοσιονομικές προσαρμογές για το 2014 και 2015 είναι κατά τη χαμηλότερες από εκείνες που είχαν συστηθεί φέτο. Είναι όμως πολύ σημαντικό σε ανταλλάγμα η Γαλλία να αξιοποιήσει αυτόν τον επιπλέον χρόνο για να ε, αντιμετωπίσει τα υποκείμενα προβλήματα οικονομικής ανταγωνιστικότητας που έχει. Για παράδειγμα, συνιστούμε στη Γαλλία να μειώσει έτσι περαιτέρω το εργασιακό κόστος, ε, μειώνοντας ε, τις συνεισφορές στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Το επιχειρηματικό περιβάλλον και η καινοτομία και η δυνατότητα εξαγωγών των εταιριών, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, θα πρέπει να ενισχυθούν. Επίσης, θα πρέπει η αγορά να ε, λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει την απασχόληση. Θα πρέπει μέχρι τέλη του έτους ε, να ε, επιληφθούν του συνταξιδοτικού συστήματος για να είναι βιώσιμο το σύστημα μέχρι το 2020. Η Ισπανία το τελευταίο έτος έχει διεξάγει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις, ε, αλλά ακόμα υποφέρει πολύ, πολύ ψηλή ανεργία και χρέος που προέκυψε μετά από ε, την ε, κρίση μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει υποβάλει η Ισπανία είναι πιστικό και εμείς τη συστήνουμε να επικεντρωθεί εκεί με τρόπο ε, αποτελεσματικό και αυστηρό. Η ε, Σλοβενία ε, αντιμετωπίζει σε βάθος τα προβλήματά της. Θα πρέπει γρήγορα να προχωρήσει και μεταξύ αυτών να αντιμετωπίσει τα ζητήματα του τραπεζικού τομέα. Οι ε, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις λοιπόν είναι κάτι που μας απασχόλησε. Οι συστάσεις είναι πιο συγκεκριμένες, πιο ε, ευκρινείς και πιο ευρείες από ό,τι στο παρελθόν. Με βάση και την πρώτερη εμπειρία μας και την καλύτερη συλλογική κατανόηση των προβλημάτων και ε, των εμποδίων στην ανάπτυξη σε διάφορες χώρες αυτό χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται μέσα σε μια τριετία που έχουμε αυτή την οικονομική διακυβέρνηση. Για να επιτύχουν οι συστάσεις μας όμως θα πρέπει να είναι αντικείμενο ευρεία συζήτηση και θα πρέπει να γίνουν κτήμα ε, της κάθε χώρας. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια έχουν εδώ να διαδραματίσουν ένα ρόλο πάρα πολύ πρωταγωνιστικό. Οι συστάσεις δεν είναι επιταγές των Βρυξελών. Ε, στη τελική ανάλυση είναι συστάσεις του Συμβουλίου και η έκφραση ε, της εταιρική σχέσης μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Εταιρική σχέση για μεταρρύθμιση, εταιρική σχέση για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Βεβαίως έχω πλήρη επίγνωση ότι είναι πολιτικά δύσκολες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ στα κράτη-μέλη, στο ΕΚΟΦΗΝ ε, κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας και να τους ζητήσω να μην αποδυναμώσουν αυτές τις συστάσεις. Ε, θα πρέπει να έχουμε την αίσθηση του κοινού ενδιαφέροντος, συμφέροντος και ανησυχία όταν σχεδιάζουμε τέτοιες οικονομικές πολιτικές και τις συζητούμε. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω το εξής. Γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρώπη ε, διασχίζει μια βαθιά οικονομική αναπροσαρμογή και μεταρρύθμιση οι μακροοικονομικές πολιτικές ε, ε, υπάρχουν για να διευκολύνουν την ανάκαμψη της οικονομίας. Η ε, νομισματική πολιτική είναι κάτι που μπορεί να προσαρμόζεται και να μεταβάλλεται. Η εξηγίαση του προϋπολογισμού έχει μειώσει τα ελλείμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τι γίνεται με τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτό θα απασχολήσει την άλλη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τώρα είναι υψή τη σημασία η ανάσα αυτή που έχει δοθεί από την επιβράδυνση λίγο των διαδικασιών ε, εξυγίανση να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη-μέλη για να κάνουν εκείνε τι μεταρρυθμίσει που χρειάζονται οπωσδήποτε για να απελευθερωθεί όλο το δυναμικό ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Σας ευχαριστώ πολύ. Βλέπουμε ότι τα, τα χειροκροτήματα δεν έλειψαν. Θα ακούσουμε τώρα τον Επίτροπο Άντορ για 10 λεπτά. Uh, Αξιότιμοι βουλευτές, πρόεδρε, στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου μου, ασχολούμε με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και βασιζόμαστε σε τέσσερα βασικά έγγραφα που συνετάχθησαν τους 16 τελευταίους μήνους για το πακέτο απασχόλησης του περασμένου Σεπτεμβρίου, το συνολικό πακέτο απασχόλησης και το ε, ε, πακέτο κοινωνικών επενδύσεων. Τώρα, οι ειδικές συστάσεις ε, βασίζονται στην προϊούσα διαδικασία που σχετίζεται με όλα αυτά τα πακέτα η Επιτροπή Απασχόλησης καθώς και η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας διαδραματίζουν κέριο ρόλο διότι εποπτεύουν τις εξελίξεις στα κράτη-μέλη και μας βοηθούν να εντοπίζουμε τις βασικές προκλήσεις ανά κράτος μέλος επί τη βάση των εργασιών των κρατών μελών για τα επιμέρους ζητήματα. Πριν περάσω στο, στις συγκεκριμένες συστάσεις, θα ήθελα να αρχίσω με μια σύσταση που συνδέεται με τη σημερινή απόφαση για τη συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης. Θα έχετε ενημερωθεί κατά πάσα πιθανότητα ότι σήμερα εγκρίνεται μια πολύ σημαντική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης στους κόλπους τη Ευρωπαϊκή Ένωσης που θα μα βοηθήσει όχι μόνο θα σπίσουμε καλύτερα πρότυπα αλλά να έχουμε και συγκρίσιμα μεγέθη ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών και ως εκ τούτου καλύτερη, καλύτερο συντονισμό των πολιτικών απασχόληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στα πλαίσια των ειδικών αναχώρασης τάσεων διότι κάποιες χώρες όπως και το Βέλγιο και η Ουγγαρία έλαβαν ειδικέ συστάσεις με τρόπο ώστε να ε, βελτιώσουν τις επιδόσεις τους ε, καθώς και τη, ε, έχοντας στόχο και την αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. Βλέπουμε λοιπόν πόσο κέριος θα είναι ο ρόλος των κρατικών αρχών κατά την υλοποίηση συγκεκριμένων προτάσεων ε, και ε, την πραγμάτωση των δεσμεύσεων που έχουμε αναλάβει για την βελτίωση της κατάστασης απασχόλησης κυρίως για πληθυσμιακές ομάδες όπως οι νέοι. Τις τελευταίες εβδομάδες ε, έχει ενταθεί ο διάλογος για την απασχόληση όχι μόνο στα θεσμικά όργανα της Ένωσης αλλά και σε επίπεδο αξιωματούχων των κρατών μελών αρμοδίων για την απασχόληση σε διάφορα επίπεδα. Η, πλέον βασική και μεγάλη πρόκληση για την Ένωση είναι η ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα παράδεκτα και ιδιαίτερα δυσθεώρητα επίπεδα ανεργίας στα κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε των νέων. Χρειαζόμαστε ειδική ε, δράση, ε, στοχευμένη δράση. Ε, επιγόντω, θα πρέπει να αναλάβουμε συγκεκριμένα βήματα. Εγγυήσεις για τους νέους, όπως συμφώνησε και το Συμβούλιο με ειδικέ διατάξεις, ούτως ώστε όλοι κάτω από τα 25 να λάβουν μία πρόταση για απασχόληση ως προς την κατάρτιση, ως προς τις πρακτικές ασκήσεις με το που ολοκληρώνουν την κατάρτιση εξάρτηση ή την εκπαίδευσή τους, ε, να ενισχύσουμε τα οικονομικά κίνητρα για την πρόσληψη των νέων στις επιχειρήσεις, σε περισσότερες πρακτικές ασκήσεις ε, και ε, μείωση του ποσοστού του νέων που εγκαταλείπουν το σχόλιο. Η μείωση της μακροχρόνιας ανεργίας στα κράτη-μέλη είναι μεγάλη απειλή για την σταθερότητα της αγοράς εργασίας. Χρειαζόμαστε καλύτερους στόχους για τους μακροχρόνια ανέργους, ούτως ώστε να υπάρχει εξειδικευμένη καθοδήγηση για τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων ε, μέσα από σεμινάρια, πρακτικές ε, ασκήσεις ε, που θα πηχούν τις ανάγκες σε κάθε αγοράς εργασίας ξεχωριστά. Η συνεργασία, στην οποία αναφέρθηκα στην εισαγωγή μου, ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες αρμόδιες για την απασχόληση, έχει ως εκ τούτου κέριο ρόλο. Ε, επίσης, ε, οι δημόσιες αυτές ε, υπηρεσίες θα πρέπει να λάβουν τις απαιτούμενες επενδύσεις, ούτως ώστε να ενταχθούν το ταχύτερο δυνατό στην αγορά εργασίας οι άνεργοι. Το πακέτο με τις ειδικέ συστάσεις τονίζει επίσης ότι στις πλεονασματικές χώρες βλέπουμε ότι έχουμε θετικά αποτελέσματα μετά από δράσεις που έχουν αναλυθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να προβληματιστούμε γενικότερα σε σχέση με τις αδυναμίες και τις ανεπάρκειες των κρατών μελών και τον αρνητικό αντίκτυπο που έχουν για την υλοποίηση στόχων. Τα εργαλεία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθούν, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο συντονισμό των πολιτικών απασχόλησης και των υπηρεσιών. Πολλές ειδικέ συστάσεις σχετίζονται με την ένδυα και κυρίως την παιδική ένδυα. Ε, θα πρέπει λοιπόν να ενισχυθούν τα κοινωνικά δίκτυα ασφαλείας, αντιμετωπίζοντας τη φτώχεια και και την αποτελεσματικότητα των σχετικών επιδομάτων και κρατικών υπηρεσιών. Δίνεται καθοδήγηση μέσα από τις συστάσεις στο κεφάλαιο επενδύσεις για τα παιδιά. Στη συνέχεια έχουμε ειδικέ συστάσεις Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία και αναφέρεται ότι έχουμε ε, πληθυσμιακές ομάδες ευάλωτες όπως η Ρωμά ε, που υφίστανται προβλήματα κοινωνικής ένταξης και διακριτική μεταχείριση ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η μεταρρύθμιση των συστημάτων υγείας και μακροχρόνιας περίθαλψης. Χρειάζεται επανεξέταση αυτό το ζήτημα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε όχι μόνο οικονομική βιωσιμότητα αλλά και κατάλληλη πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες και βελτιωμένη κάλυψη για το γυράσκοντα πληθυσμό της Ένωσης. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε το, τα συστήματα υγείας προς το κόστος τους και την αποτελεσματικότητά τους θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και στην ανεξάρτητη ζωή. Τέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει κάποια από τα μέτρα αυτά πολιτικής που αναφέρθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ε, ξέρετε πολύ καλά ότι από την συνθήκη έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, καθώς ε, και το σύστημα για την εγγύηση για την νεολαία. Επίσης, το πακέτο κοινωνικών επενδύσεων ε, θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προωθήσουν τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, ούτως ώστε να δώσουν μεγαλύτερη κοινωνική υποστήριξη στον πληθυσμό τους. Ε, έχουμε λοιπόν την πρωτοβουλία για την νεολαία, το, τη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ακόμα συνεχίζονται και επομένως πολλές από τις σημαντικές λεπτομέρειες ε, συζητώνται ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και στα κράτη-μέλη. Αυτά και ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Και τώρα θα περάσουμε στον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Θα ακούσουμε για τρία λεπτά τους εισηγητές ε, της ΕΚΟΝ και της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και πέντε λεπτά απαντήσεις από τον Επίτροπο ή Επιτρόπους. Η Ελίζα Φερέιρα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροποι, σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. Αυτή τη στιγμή έχουμε περιέλθει με κατάσταση όπου είναι δυνατόν να κάνουμε έναν απολογισμό των αποτελεσμάτων των πολιτικών που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τούδε. Τρόπον επικροτώ την ύπαρξη ειδικών συστάσεων για τις ανισορροπίες που υπάρχουν στην Ευρωζώνη, διότι πιστεύω ότι με τη μέθοδο ανάλυση των υπερβολικών ελλημάτων ε, σε διακρατικό επίπεδο και όχι μόνο στο εσωτερικό κάθε κράτος μας δίνει το απαιτούμενο περιθώριο αναπροσαρμογής για τα δημόσια ελλείμματα και τα δημόσια χρέη. Τούτου λεχθέντος θα ήθελα ανοιχτά να θέσω κάποια ερωτήματα προ είδαμε τον πρόεδρο της Γαλλίας ε, να αποστασιοποιείται κατά κάποιο τρόπο από τις συστάσεις. Σήμερα ο Μπερλουσκόνη ξεκάθαρα ε, παρακινεί την κυβέρνηση να μην συμμορφωθεί με το στόχο του 3% για το έλλειμμα, διότι βάσει των πληροφοριών του τύπου φέρεται να λέει ε, ο Μπερλουσκόνη ότι δεν θα εκδιωχθεί η Ιταλία από την, από την Ευρωζώνη. Στην Ισπανία έχουμε τις βασικές ε, πολιτικές δυνάμεις ε, της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά της πολιτικής λιτότητας. Και ρωτώ το εξής, όταν η κρίση πλήττει τις ισχυρότερες χώρες, τις σημαντικότερες χώρες τι συμβαίνει με τα μέτρα σε σχέση με το BRICS, ε, με την ε, Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία. Δεν θα έπρεπε να αναρωτηθούμε ε, για την ποιότητα των προγραμμάτων. Μήπως τώρα έχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε να κάνουμε μια σταθμισμένη προσαρμογή με τρόπο ώστε να λάβουμε υπόψη οικονομικές συνθήκες που ισχύουν. Ε, βλέπουμε επίση τις δηλώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα ε, και διαβλέπουμε μία πελώρια δυσκολία στην Κύπρο παραδείγματο χάρη για να αποδεθούν ευθύνες για τα μέτρα. Σας δίνω δύο-τρία συγκεκριμένα παραδείγματα απλώς. Ε, Λοιπόν, ε, ε, ρωτώ, ε, με μία πιο σφαιρική προσέγγιση του ζητήματος και ενώπιση του επομένου Συμβουλίου, μήπως θα έπρεπε να αντικαταστήσουμε την Τρόικα με μία ευρωπαϊκή μέθοδο που θα συνοδεύει αυτές τις χώρες στη διαδικασία προσαρμογής, μία, έναν εξευρωπαϊσμό του ESM, του Μηχανισμού Σταθερότητας, παραδείγματος χαρή, όπως είδαμε και σε ε, παρελθούσες περιόδους ότι υπάρχουν άλλες δυνατότητες ε, δράσης. Ε, μήπως θα έπρεπε να ασχοληθούμε με το, την ομάδα που θα ασχοληθεί με το ειδικό Ταμείο Διάσωσης όπως επίσης μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έχουμε ένα νέο εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα και τι γίνεται με τις επενδύσεις που θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε ούτως ώστε με προληπτικό τρόπο να αποφύγουμε τα υπερβολικά ελλείμματα, επιτρέποντας όμως ε, ε, την ανάπτυξη, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να αντικαταπολεμήσουμε την ε, ανεργία. Ευχαριστούμε, Λίζα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο για τους εισηγητές. Αλλά... πρέπει να μιλάμε λίγο πιο λακωνικά. Βερόνικα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Λόπε. Ευχαριστώ και τους επιτρόπους. Ε, που ήρθαν εδώ στις δύο επιτροπές μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα να ευθυγραμμίσουμε και να συντονίσουμε την οικονομική και την κοινωνική πολιτική ε, και να πούμε από την κρίση. Εγώ θα περιοριστώ στο τρίλεπτο, Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια έκθεση για την απασχόληση που επικέντρωνε σε κάποια σημεία κλειδιά για τις συστάσεις αναχώρα. Το πρώτον, είπαμε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η εφαρμογή των απαραίτητων εκείνων μέτρων για να πλησιάσουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020 και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απασχόληση και τη μείωση της ένδυας. Ορισμένες χώρες ήδη τα υλοποιούν αυτά. Ε, άλλο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και ο Επίτροπος Ρεν, αλλά δεν θα επεκταθώ γιατί θεωρώ ότι συμφωνούμε όλοι, είναι ε, η ισορροπία ανάμεσα στην εξυγίανση των προϋπολογισμών και την κοινωνική πολιτική. Αυτή η ισορροπία παραμένει για μας προτεραιότητα. Αλλά θα ήθελα εδώ να διαφωνήσω λίγο με την ε, ε, σοσιαλίστρια συνάδελφο της Οικονομικής Επιτροπής. στη συμφωνία του ε, Λαϊκού Κόμματος με το Σοσιαλιστικό στην Ισπανία στόχος δεν είναι ε, να τερματιστεί η, η ε, λιτότητα, αλλά να προωθηθούν θέματα απασχόλησης και μάλιστα ποιοτική απασχόλησης για χώρες όπως η δικιά μου. Αυτό θα πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθούν τα ενεργά μέτρα της εργασίας όπως υπηρεσίες κατάρτισης και απασχόλησης για να μην ε, φεύγει νωρίς ε, από την αγορά από το σχολείο νέος. Και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, αν θέλουμε να είναι ο κινητήρας της απασχόλησης, θα πρέπει να τις βοηθήσουμε και να τις βοηθήσουμε στη χρηματοδότησή τους, στη δανειοδότηση και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων. Και τελειώνω με πολλές ερωτήσεις που έχω προς τους επιτρόπους. Εδώ και πολύ χρόνο ακούμε για την εγγύηση για την νεολαία, αλλά τελικά ο απαραίτητο προπολογισμό λέει θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να είναι εμπροσοβαρές αυτό το πρόγραμμα γιατί είναι απαραίτητο για κάποια κράτη-μέλη. Δεύτερο, ε, τι γίνεται με την ε, επιταχυμένη ε, εγγραφή και απορρόφηση των 16 δισεκατομμυρίων για τους νέους. Τρίτον, για τον κατακαιρματισμό των χρηματαγορών. Αυτό έχει να κάνει ε, με την απασχόληση. Θα καταφέρουμε επιτέλους μια τραπεζική ένωση για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δανειοδοτούνται με ε, το ίδιο επιτόκιο και τους ίδιους όρους ανεξαρτήτως έδρας. Ευχαριστώ. κάθε επίτροπος έχει πέντε λεφτά. Όλοι πρώτος. Ευχαριστώ Σάρον. Ευχαριστώ και τους δύο εισηγητές ή εισηγήτρες καλύτερα, για τα σχόλια και ερωτήσεις. Κυρία Φερέιρα, καταρχήν, είπε κάποια πράγματα αναφερόμενοι σε δηλώσεις πολιτικών ηγετών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστό να πούμε, είναι να πούμε ότι η μεταρρύθμιση της ε, Ευρώπης είναι μεγάλη πρόκληση και η πολιτική συζήτηση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων και αυτές στις οποίες αναφερθήκατε, ακριβώς απεικονίζει αυτή η δυσκολία και το βαθμό της πρόκλησης που είναι και οικονομική και πολιτική που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Οι συστάσεις μας βασίζονται σε μια οικονομική ανάλυση. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη σε μια εταιρική σχέση μαζί τους για να μεταρρυθμίσουν τις κοινωνίες τους και να μπορέσουν να απελευθερώσουν το δυναμικό που έχουν για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και περιμένω τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο να επικυρώσουν τα σχέδια συστάσεων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για τα 27 κράτη, μεταξύ των οποίων και αυτά που αναφερθήκατε στις παρατηρήσεις σας, κυρία Φερέιρο. Αυτό συνδέεται τώρα και με την ερώτησή σας για τα μεγάλα και τα μικρά κράτη. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ίση μεταχείριση των κρατών μελών. Θέλω να αναφερθώ ιδίως στην περίπτωση της Γαλλίας, που συχνά χρησιμοποιείται ως παράδειγμα. Συστήσαμε επέκταση δύο ετών αντί για ενός έτους στη Γαλλία για την ε, εξυγίαση των δημοσίων οικονομικών. Γιατί γιατί κάναμε μια οικονομική ανάλυση που έδειξε ότι αυτός είναι καλύτερος τρόπος για να μπορέσει η Γαλλία και η Ευρωζώνη να προχωρήσει. Η Γαλλία θέλει να φέρει το ή ήθελε τουλάχιστον αριστερά αρχικά να φέρει το έλλειμμα κάτω από το 3% του χρόνου. Και θα ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό με διαρθωτικούς όρους μέχρι το 2016. Η Κομισιόν πιστεύει ότι αυτό είναι υπερβολικά αισιόδοξο και η δημοσιονομική προσπάθεια που προβλέπουν οι αρχές δεν συνάδει με την ε, σημερινή διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος που θα λάβει η χώρα μέχρι του χρόνου. Εκτός και αν ληφθούν και άλλα μέτρα για να αντισταθμίσουμε αυτό που θεωρούμε εμείς υπερβολικά αισιόδοξο μακροοικονομικό σενάριο. Η επιπλέον προσπάθεια που χρειάζεται για να κατέβει το έλλειμμα κάτω το 3% του ΑΕΠ και η επίπτωση που η περαιτέρω εξυγίανση θα είχε στην ε, οικονομική ανάπτυξη βράχη πρόθεσμα, ανάγκασε την Κομισιόν με βάση την οικονομική ανάλυση που κάναμε να προτείνουμε την επέκταση της προθεσμίας σε δύο χρόνια αντί για ένα χρόνο, αντί για, ένα χρόνο για τη Γαλλία, ούτως ώστε να διορθώσει τα, τις υπερβολές, το υπερβολικό έλλειμμα μέχρι το 2015 το αργότερο. Είναι πολύ σημαντικό η Γαλλία να χρησιμοποιήσει αυτό το χρόνο που της δίδεται, ούτω ώστε να προβεί στις διαφορετικές ε, μεταρρυθμίσεις ε, στο σύστημα συντάξεων, στην αγορά εργασίας, ούτω ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική η γαλλική οικονομία και πιο ικανή να δημιουργεί θέσει απασχόλησης. Ρωτήσατε λοιπόν επίσης για τη λειτουργία της Τρόικα και τη δυνατότητα εξευρωπαϊσμού των δράσεων σταθερότητας. Να σας υπενθυμίσω ότι οι αποφάσεις μας να δημιουργήσουμε το σημερινό μοντέλο, αυτό που ονομάζουμε Τρόικα, δηλαδή Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Δούνου του, αυτή την απόφαση την έλαβαν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης την άνοιξη του 2010. Και πολλά κρατημέλη επέμειναν να μπει και το δούνου του στην Τρόικα. Δουλέψαμε μετά από αυτή την εντολή που μας δώσαν τα κρατη της Ευρωζώνης. Σε ό,τι αφορά τα σημερινά προγράμματα. Και θα συζητήσουμε τους καλύτερους και βέλτιστους τρόπους για να προχωρήσουμε και στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια ευρύτερη συζήτηση για την ε, αναδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής και Νομισματικής ε, Ένωσης. Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Επίσης, τι ε, δράση σταθερότητας πρέπει να προωθήσουμε όταν μια χώρα αντιμετωπίζει υπερβολικές δυσκολίες. Ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, αλλά η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη μερική έκδοση χρέους στην Ευρώπη και τα ευρωομόλογα, αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων είναι στην τελική φάση των εργασιών της, θα κάνει προτάσεις και πιστεύω ότι στις επόμενες 15 μέρες θα είμαστε σε θέση να έχουμε τις προτάσεις της ομάδας αυτής, ούτως ώστε η Επιτροπή μετά από αυτές τις προτάσεις να αρχίσει τη δουλειά της πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. με τις εγγυησει των νέων, Έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες, εκ των οποίων η πιο σημαντική είναι οι εγγυήσεις για τους νέους. Τραβούν όλο ένα και περισσότερο την προσοχή. Είδατε, Ε, την ε, συνάντηση υψηλού επίπεδου που άρχισε στο Παρίσι και συνέχισε την περασμένη εβδομάδα στη Ρώμη και αυτή τη βδομάδα στη Μαδρίτη και θα τελειώσει στο Βερολίνο κατά πάσα πιθανότητα την 3η Ιουλίου. Ε, προβάλλεται δηλαδή ε, το νέο μέτρο και πολλοί πλήττονται από την κρίση και κυρίως από την ανεργία των νέων. Ε, και έπρεπε να συνεννοηθούμε ούτω ώστε ε, από, τον υπερβολικό αριθμό μεών να μην χάσουμε το παιδί του στο τέλος. Πρέπει οι δράσεις μας να ανταποκρίνονται στις ε, απαιτήσει ε, των ανέργων ε, και να εκμεταλλευτούμε τον νέο αυτό ενθουσιασμό που επικράτει. Βεβαίως διαπιστώνονται αναμφίβολα ανεπάρκειες. Η πρωτοβουλία για τους νέους προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. 6 δις ήταν το κονδύλι το Φεβρουάριο. Ε, τώρα οδεύουμε προς μια συνένεση ότι θα πρέπει να είναι έμπροστο βαρύς η εκταμείευση του κονδυλίου για την προβλεπόμενη περίοδο. Δεν είναι πλήρης η συνένεση, ε, ε, εκκρεμούν κάποια τεχνικά ζητήματα, όμως πολιτικός και οικονομικός πώς είναι πολύ λογική αυτή η πρωτοβουλία. Τα έξι αυτά δις θα πρέπει να θεωρηθούν ως προσάυξηση, top Ορισμένες φορές εικάζουν κάποιοι ότι δεν θα υπάρξει άλλο κονδύλι για την πρωτοβουλία για τους νέους. Ε, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ε, ως επιτοπλίστων ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα είναι η πηγή χρηματοδότησης για τέτοιου είδους ε, δράσεις ε, και είναι πολύ λογικό το νέο εργαλείο να συνειδητοποιήσουμε ότι θα δώσει μια χρηματοδότηση εν είδη σε συγκεκριμένες περιοχές και το ποσοστό θα πρέπει να είναι άνω του 25%. Μετά τη συμφωνία του Συμβουλίου το Φεβρουάριο άρχισαν οι πρακτικές προεργασίες και ε, σε χώρες όπως η Ισπανία βλέπουμε αρκετά δυσεπίλητα προβλήματα ε, για το κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή του συστήματος. Ε, φυσικά το θέμα μας απασχολεί κυρίως σε σχέση με την Ισπανία και την Ελλάδα. Εάν το πακέτο αυτό διοχετευτεί ούτω ώστε να συμπεριληφθούν κονδύλια ε, από την πρωτοβουλία για τους νέους αλλά και από το ΕΚΤ για αυτές τις δύο χώρες ε, είναι δυνατόν ε, να φανταστεί κανείς ότι θα έχουμε τα απαιτούμενα κονδύλια για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα για τις εγγυήσεις των νέων. Στην Ισπανία το Μαδρίτη ε, συζητήθηκε το θέμα το Μάιο και την επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί στην Αθήνα ε, ως προς τα κονδύλια της τωρινής περίοδου 16 ε, δισεκατομμύρια ευρώ στοχεύουμε 8 κράτη-μέλη και μισό εκατομμύριο νέους εκεί όπου παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συνολικό ποσό θα ήταν 5,1 εκατομμύρια. Ταυτόχρονα ε, επιδεινώθηκε η ύφεση και στο ενδιάμεσο διάστημα αυξήθηκε ο αριθμός των ανέργων νέων και ο καθαρός αντίκτυπος αυτών των κονδυλίων δεν είναι τόσο μεγάλος όσο περιμέναμε και θα επιδεινωθεί η κατάσταση όσο επιδεινώνεται και η ύφεση. Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα εγγυήσεων για τους νέους. Ε, είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και να έχει απτά αποτελέσματα ε, χρησιμοποιώντας τα τωρινά, ε, τους τωρινούς μηχανισμούς και γι' αυτό ταυτόχρονα ε, επιδιώκουμε και άλλους στόχους εκ για να τονώσουμε την απασχόληση αλλά και εν γέννη την οικονομική μεγέθυνση. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωταπαντήσεων. Δύο λεπτά έκαστος για τους διαφόρους ομιλητές. Guterres, Prieto, Niels Torvalds and uh, Pablo uh, Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Αλπαμπιδεγάιν. Ε, μία από τις προτεραιότητες ε, στην ε, έκθεση ε, για την αιτήσια ανάπτυξη ήταν να επανέλθει η ε, φυσιολογική πίστη ε, στην οικονομία. Ήταν η έκθεση της κυρίας Λόπε Φοντανιέ. Είναι σημαντικό να χρηματοδοτούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι με βάση την έδρα της εταιρείας αλλά με βάση την κατάσταση. Ήδη από το 2012 στην αιτήσια αυτή η έκθεση για την ανάπτυξη ήταν προτεραιότητα αυτό το ζήτημα και η κατάσταση δεν έχει σταματήσει να επιδεινώνεται ε, στις χώρες του Νότου, όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία. Στις χώρες αυτές οι μικρομεσαίες χρηματοδοτούνται μέχρι και 70% ακριβότερα από τις άλλες χώρες. Και μάλιστα πέρσι στην Ισπανία έπεσαν τα δάνεια για τις μικρομεσαίες ε, κατά 23 και πλέον τις 100. Χωρίς τις μικρομεσαίες όμως δεν πρόκειται να έρθει ανάκαμψη στην οικονομία. Και επιπλέον η κρίση στο πρόβλημα αυτό είναι εξόχως ευρωπαϊκή. Εντάξει, ο ενιαίος επόπτης ε, θα αρχίσει να μπλέκει αυτές τις ε, αγορές, αλλά μέχρι τότε δεν πρόκειται να λυθεί η κατάσταση. Λοιπόν, κύριε Επίτροπε Ρεν, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο ε, για να βελτιωθεί η κατάσταση, πόσο μάλλον που αυτό το θέμα είναι προτεραιότητα από το 2012. Και θα ήθελα και στον κύριο Άντορ να πω ότι χαίρομαι για τον ενθουσιασμό του. Λέει ότι η προτεραιότητά του είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και δι των νέων στην Ευρώπη. Μάλιστα. Αλλά δεν θα πρέπει όμως να ε, κοιτάμε και πιο μακροπρόθεσμα τι γίνεται και να δούμε στρατηγικές πώς θα μπορέσουμε στο μέλλον επίσης να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που είναι και σοβαρά και μεγάλα της ανεργίας. Λοιπόν, συμφωνούμε στη διάγνωση. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε ότι η λύση είναι περισσότερη Ευρώπη για την κρίση. Εσείς λοιπόν κύριε Επίτροπε πώς θα αξιολογούσατε στο μέλλον μια ενδεχόμενη μερική έστω συνένωση ε, του συστήματος ε, ε, ασφάλισης κατά της ανεργίας. Ευχαριστώ. Ο Σέργιο. Σέργιο, κύριε Ρεν, τόσο πολύ απέχουμε από τις συστάσεις σας ε, και όχι μόνο γεωγραφικά, πόσο απέχουμε εδώ από το πάνελ. Πριν από λίγους μήνες είχατε έρθει εδώ και συζητήσαμε την ετήσια έκθεση για έρευνα για την ε, ανάπτυξη. Ε, σας είπαμε ότι η υπερβολική λιτότητα επηρεάζει πάρα πολύ την καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών. Και από τότε με πολύ μεγάλο σθένος ε, αρνηθήκατε τα θέματα των ε, πολλαπλασιαστών και μιλούσατε για τήρηση του προγράμματος. Μα όλοι οι πάντες μας έλεγαν το δουνού του, οικονομικά Ινστιτούτα, όλοι ομολογούν το λάθος τους και εσείς οι ίδιοι. Παρ' όλα αυτά ε, συνεχίζετε να μας παρουσιάζετε την ίδια στρατηγική. Κύριε Επίτροπε, πιστεύετε ότι θα σας χειροκροτήσει και από πάνω η σοσιαλιστική ομάδα επειδή μας δώσατε δύο χρόνια παραπάνω για ορισμένα κράτη-μέλη ή Είπατε στη Γερμανία να αυξήσει λίγο τους μισθούς για να τονώσει την εσωτερική ζήτηση, βασικά μειώνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές. Μα χρειαζόμαστε πιο βαθιά αλλαγή στρατηγική για να βγει από την κρίση Ευρώπη. Όχι καλοπιστικές πολιτικές ε, για να μακιγιάρουν την αποτυχία σας ε, ε, που δεν μπορείτε να βγείτε από την κρίση. Λοιπόν, Πώς δικαιολογείται ότι παρά την προθεσμία των δύο απαιτείται από κάποιες χώρες να μειώσουν το ΑΕΠ δύο και τρεις φορές πιο ε, περισσότερο από ό,τι ε, είχαμε συμφωνήσει στο six pack. Μια μελέτη ε, που ζητάει αντικειμενικό χρονοδιάγραμμα και όχι υποκειμενικό, πολιτικά κινούμενο και αλακάρτ όπως κάνετε εσείς. 0,7% στην Ευρωζώνη μπορεί ετησίως να τονωθεί ε, το ΑΕΠ. Θα μπορούσατε να μου πείτε πόσους πόρους χάσαμε, πόσους ε, ανθρώπους που έμειναν ε, από επίδομα ανεργίας, που έμειναν από υποτροφία μπορείτε να τα προβλέψετε όλα αυτά οικονομικά. Γνωρίζετε ότι από τις τελευταίες 13 προβλέψεις σας οι 11 έπεσαν έξω κατά μισή ποσοστιαία μονάδα τουλάχιστον. Με αυτές τις παραβέντρους μήπως πρέπει να αλλάξετε υπολογιστές ή φόρμουλες. Μα είναι ασυνάρτητα αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν από τη μια ε, εκφράζει τη λύπη της για τη μείωση ε, των πόρων στην υγεία, στην παιδεία, αλλά μετά όταν σας φέρνουν τα εθνικά σχέδια, τα κράτη-μέλη, δεν λέτε τίποτα. Συγγνώμη, πρέπει να σας ε, διακόψω. Να έρχεται πιο συχνά ο Επίτροπος για να του τα λέμε, να τα ακούει από τους σοσιαλιστές. I, I, I... Καταλαβαίνω ότι έχετε να πείτε πολλά, αλλά υπάρχουν και πολλοί που θέλουν να πάρουν το λόγο όμως και, που και αυτοί θέλουν να πούν πολλά. Ο Νίλς είναι ο επόμενος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπάμαι για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται συνήθως η συζήτηση εδώ στην Επιτροπή Εκόνα. Μακάρι να ήταν ο Όλι Ρεν ε, στην ε, επικεφαλής ας πούμε, της κυβερνής της Ελλάδας, της Ισπανίας, ε, ε, της Ιταλίας, αλλά δεν ήταν όμως επικεφαλής. Τι να κάνουμε. Για τις οικονομικές σας αναλύσεις. Μας έχετε μιλήσει πολύ για αυτές. Όταν όμως βλέπουμε την ε, πραγματικότητα και τη θεωρία, βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Υπάρχει η καμπύλη Φίλιπς Πολλοί οικονομολόγοι τη χρησιμοποίησαν ως μαθηματική βάση μετά την ύφεση. Βλέπετε αυτή την θεωρία. η οποία μας στέλνει στα βάραθρα. Ειδικά όταν συζητάμε με το Δουνουτού. Αυτή η θεωρία της κατακαιρμάτισης, πόσο επηρεάζει τη σκέψη σας. Πώς μπορείτε με αυτή τη θεωρία να κάνετε καλή δουλειά, τέλος πάντων. Κυρία Um, thank you Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που ήρθατε και οι δύο. Ευχαριστώ και τους δύο επιτρόπους. Θέλω να σας ρωτήσω για την πρόοδο που κάνατε στα σχέδιά σας για να ενισχύσετε την ε, κοινωνική διάσταση Τον Απρίλιο η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών είχατε πει ότι θα αναπτυχθεί περαιτέρω. Ο κύριος Άντορ μίλησε για το πίνακα επιδόσεων για τις ε, μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ε, δεν, έχει όμως, ε, δεν υπάρχει πια τέτοιος πίνακας. Δεν έχει, τον περιμένουμε αλλά δεν έχει, μας έχει δοθεί. Οι κοινωνικές ανισορροπίες, όπως η υπερβολική ανεργία των νέων, αύξηση του επίπεδου φτώχειας, η αύξηση των ανισοτήτων, πόσο θα είναι αποφασιστικές στις μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών. Και πώς θα λυθούν υπόψη ε, από την Επιτροπή. Ε, στα πλαίσια της διαδικασίας υπερβολικού ε, ελλείμματο και υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Θα κάνετε σχετικέ προτάσει ή τι περιμένουμε για το επόμενο εξάμενο. Δεν έχω πολύ χρόνο. Θα ήθελα να σα ρωτήσω και κάτι άλλο για την εμπλοκή τη κοινωνία των πολιτών. Πρέπει να ομολογήσετε τα τελευταία χρόνια η δημόσια στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης δεν, δεν ήταν πολύ λαμπρή. Και υπάρχουν πολλές ανησυχίες για τη δημοκρατική διαδικασία. η κοινωνία των πολιτών εκπροσωπεί εκατομμύρια Ευρωπαίους, αλλά δεν ακούεται επαρκώς τη διαδικασία που εφαρμόζεται. Υπάρχουν κάποια σχέδια για να βελτιώσετε την... υπάρχειτε περίπτωση, υπάρχει περίπτωση να δώσετε φωνή και σε αυτούς τους φορείς, σε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Όλοι τώρα θα απαντήσει. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με την άμεση και πολύ σημαντική ερώτηση που έθεσε ο Ισπανός ομιλητής για την αποκατάσταση της, ε, του φυσιολογικού δανεισμού στην πραγματική οικονομία. Ο οικονομικός κατακαιρματισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμποδίζει την ανάπτυξη, συμφωνώ και ίσως είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που παρεμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη. Αν λάβουμε υπόψη μας ειδικά την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Νότια Ευρώπη, σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία. Είναι σημαντικό να συμπληρώσουμε τη δουλειά της οικονομικής ανάκαμψης, της δημιουργίας της Τραπεζικής Ένωσης, με συγκεκριμένε πρωτοβουλίε πολιτικής, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της ε, χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Που, που έχει πρόβλημα πραγματικά α, ρευστότητας. Τι πρέπει να κάνουμε. Να δούμε τους ισολογισμούς των τραπεζών, να τους στηρίξουμε, ούτως ώστε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό το να γίνει μια αξιόπιστη αξιολόγηση της Ευρωζώνης, των τραπεζών της Ευρωζώνης, που θα γίνει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Εποπτείας, κάθετος Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και από τις δύο δηλαδή, μαζί με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Είναι σημαντικό, επίσης, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να κάνουν ό,τι μπορούν, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα της χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και γι' αυτό η Κομισιόν συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ούτω ώστε να βρούμε ένα σύστημα που θα δίνει γρήγορη βοήθεια Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα δώσει την πρώτη εγγύηση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με βάση την εντολή που έχει και με ανεξάρτητη απόφαση θα βοηθήσει για να αυξήσει τον όγκο αυτού του συστήματος, του σχήματος εμπασπιπτώσεων, ώστε να έχει πραγματική επίπτωση η προσπάθεια αυτή στην πραγματική οικονομία της Ευρώπης. Ολοκληρώνουμε μία έκθεση και μία πρόταση για αυτό το θέμα στο εσωτερικό της Κομισιόν μαζί με την ε, ΕΚΤΑ και ελπίζουμε να ετοιμάσουμε αυτή την πρωτοβουλία πριν από την ε, Σύνοδο Κορυφή ε, που θα λάβει η χώρα την επόμενη εβδομάδα. Είναι σημαντικό ε, η Σύνοδο Κορυφή να δώσει στήριξη σε αυτή την κοινή πρωτοβουλία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν απτά αποτελέσματα για τη μείωση του κόστου δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επομένω να υπάρξει ρευστότητα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει στην Ευρώπη. Ο κύριος Κουτιέρες Πιέτρο αναφέρθηκε στις συστάσεις μου και στις συστάσεις του Άντορ. Αυτές οι συστάσεις αναχώρα υιοθετήθηκαν και παρουσιάστηκαν στις 29 Μαΐου και είναι οι συστάσεις ολόκληρης της Επιτροπής, ολόκληρου του σώματος επιτρόπων που υιοθετήθηκαν ομόφωνα. Είναι προϊόν συλλογικής και σκληρής δουλειάς ε, των υπηρεσιών της Επιτροπής και των Επιτρόπων και των Γραφείων των Επιτρόπων. Και υποστηρίζω και υπερασπίζομαι αυτές τις συστάσεις στον τομέα της ε, πολιτικής ε, απασχόλησης που ετοίμασε ο φίλος μου Άντορ και φαντάζομαι ότι και εκείνος και οι υπόλοιποι θα στηρίξουν τις δικές μου συστάσεις για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και την οικονομική πολιτική. Ένα άλλο ευρωβουλευτή, όπως και ο κ. αναφέρθηκαν στις οικονομικές μελέτες και στις οικονομικές θεωρίες και αναλύσεις. Οι οικονομικές θεωρίες είναι πολύ διαφορετικέ. Υπάρχει ένα τρομερό κατακαιρματισμό. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Στην ε, Κομισιόν εμεί δεν βασιζόμαστε σε μία συγκεκριμένη μελέτη, σε, μία, σε ένα δόγμα. Κοιτάμε και βασιζόμαστε σε πολλές οικονομικές μελέτες. Και μπορώ να συνεχίσω να, να σας απαντώ σε αυτό το θέμα στον επόμενο γύρο ερωτήσεων, γιατί νομίζω ότι θα επανέλθουν κάποιοι άλλοι ενδεχομένω ευρωβουλευτέ σε αυτό το θέμα. Επομένω, θα συνεχίσω να σα απαντώ στον επόμενο γύρο απαντήσεων. Δύο λόγια. Σε σχέση με την ανεργία των νέων, ακούσαμε ερωτήσει, παραδείγματο χάρη ε, σε σχέση με την μακροπρόθεσμη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Κοιτάξτε, έχει δύο σκέλη η απάντησή μου στον τομέα της απασχόλησης και της αγορά εργασίας, ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι αλλαγές που γίνονται υπό την σκέπη της νέας πρωτοβουλίας ε, για τις εγγύσει για τους νέους αλλά και για την επαγγελματική κατάρτιση σε ορισμένες χώρες και τόνωση της κινητικότητας όπου παρατηρούνται ελλείψεις και διάφορα άλλα μέτρα θα βελτιώσουν εν γέννη το δυναμικό τους ώστε να είναι πιο ανθεκτικό το σύστημα στην αγορά εργασίας ε, και να γίνεται καλύτερα η μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας στην Ισπανία και σε άλλες χώρες ε, θα πρέπει ε, να επανεξετάσουμε το θέμα των περίφημων συμβάσεων ε, ούτως ώστε να βρούμε λύσεις για να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό της αγορα σε αυτές τις χώρες. Ε, βεβαίως το άλλο σκέλος ε, έχει ιδιαίτερη σημασία, η νομισματική ένωση η ίδια. Από ό,τι φαίνεται από την εμπειρία των περασμένων ετών βλέπουμε ότι είμαστε υπερβολικά εκτεθειμένοι σε ένα μηχανισμό boom και bust. Ε, ε, boom δηλαδή οικονομική άνθηση και bust ύφεση, οικονομική ύφεση και κυρίως εντοπίζουμε μια έλλειψη ε, σταθεροποιητών, ούτως ώστε να ανακάμπτουμε ταχύτερα όταν είμαστε σε ύφεσιακό κύκλο. Θα πρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε περαιτέρω τις λύσεις μας ε, όχι μόνο στην Επιτροπή αλλά και σε άλλα θεσμικά όργανα ώστε να είναι γνήσια και αυθεντική η νομισματική ένωση. Κυρία Κορνέλησεν, ε, μας ερωτήσατε για την για την δήλωση του Προέδρου ε, την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Πολύ σημαντική αυτή η διάσταση της αναδιάρθρωσης της ε, ΟΝΕ. Το χρονοδιάγραμμα φυσικά θα πρέπει να ε, γίνει σε συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εμείς προβλέψαμε τα πάντα σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Εάν γίνουν αλλαγές, γιατί με ενημέρωσαν ότι άλλαξαν ημερομηνίε του ΕΠΣΚΟ Συμβουλίου ε, που είχε προβλεφθεί για αυτή την εβδομάδα ε, εξυπακούεται ότι θα προσαρμόσουμε και εμείς το δικό μας χρονοδιάχρημα ε, για τις δικές μας προεργασίες. Όμως, ταυτόχρονα αληθεύει ότι το έγγραφο για την κοινωνική διάσταση καλύπτει αυτό που μας είπε ο κύριος Τούρβαλτς για τον κατακαιρματισμό. Στη συνέχεια, μιλήσατε για μια πιθανή ασφάλεια ανεργία σε επίπεδο ε, ο, ε, οι ατέλειες, οι ανεπάρκειες του τωρινού ε, μοντέλου ένωσης προϋποθέτουν διεξοδικότερη ανάλυση ούτως ώστε να αντικαταστήσουμε τους σταθεροποιητές χρέους τουλάχιστον εν μέρη σε εθνικό επίπεδο και εν μέρη ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ε, και διυπηρεσιακά στο επιτελείο του Όλη Ρεν και το δικό μου κάνουμε ήδη προσαρμογές στο προσχέδιο της επόμενης πρότασής μας και αξίζει την προσοχή μας και κυρίως ενδελεχή συζήτηση το θέμα ε, και εδώ στο Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα είναι ε, το ταχύτερο δυνατό, μου απαντάει η Πρόεδρος, το ταχύτερο δυνατό θα γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Και τώρα ήρθε η ώρα να παραδώσω την Προεδρία στην Περβάνς. Αλλιώς θα έχουμε προβλήματα χρόνου. Ευχαριστώ πολύ Σάρων, αγαπητοί συνάδελφε. Τρίτος γύρος λοιπόν ερωτήσεων από την οικονομική και νομισματική εξ των, πρασιν... των πρασίνων, λέει η πρόεδρος, ο κύριος Γιάνν Έπινγκ. Μετά ο κύριος Τούσας από την Επιτροπή Επασχόλησης. Ο κύριος Έπινγκ είναι συντηρητικός λίγο. E ah. e Α, ECR. Α, κατάλαβα ότι έτσι κάπω αναστατωθήκατε. Ε, όχι πράσινη. Λοιπόν, ECR, μετά ο κύριο Τουσα από την Επιτροπή Απασχόλησης, μετά Econ Giggold. Ε, ε, να αλλάξει λοιπόν οι επιτροπές. Ο κύριος Έπινγκ, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εντάξει, δεν κάνει τίποτα. Σας συγχωρώ. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Επίτροπο Άντορ που έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung στις 29 Απριλίου. Το διάβασα στα γερμανικά το κείμενο και λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στη Γερμανία να αυξήσει τους μισθούς για να ε, ε, τονωθεί η εσωτερική ζήτηση και να έχει ε, έναν κατώτατο μισθό σε ευρύ πλαίσιο. Εσείς εδώ αντανακλάτε τη θέση την επίσημη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Σώματος των Επιτρόπων. Αν ναι, Τότε κύριε Ρεν, γιατί δεν το έχετε βάλει αυτό ε, στις του 2013 για τη Γερμανία. Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στα δύο. Ε, τι φρονεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα. Ποια είναι η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Άντορ εξέφραζε προσωπικές απόψεις ή ε, του συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή Απασχόλησης, ο κύριος Τούσας παρακαλώ. Η παράδειση της δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν αποτελεί αλλαγή της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιτάχυση των καπιταλιστικών αναδιαθρώσεων αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κυβερνήσεων στα κράτη-μέλη της για την ενίσχυση της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Μαζική ανεργία, φτώχεια, απόλυτη εξαθλίωση. Στην κλίνη του Προκρούστη έχουν μπει οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι κλαδικές συμβάσεις, τα δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, οι δημόσιες υπηρεσίες παροχής υγείας, πρόνοιας, παιδείας. Με την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που είναι μέρος του συνολικού πακέτου της οικονομικής διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση, επιχειρείτε να φορτώσετε στους λαϊκούς ώμους το κόστος διάσωσης των τραπεζών, να βάλετε στο χέρι ακόμα το μόχθο της δουλειάς ολόκληρης ζωής. Τις πενιχρές αποταμιεύσεις όσες έχουν απομείνει, όσων λαϊκών οικογενειών κατόρθωσαν τα προηγούμενα χρόνια να βάλουν κάτι στην άκρη για την ώρα ανάγκης. Λιτότητα και αυταρχισμός αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και με αυτό τελειώνω, είναι η πρόσφατη επέσχυντη απόφαση της τρικοματικής κυβέρνησης στην Ελλάδα να κλείσει τη δημόσια τηλεόραση και να απολύσει 2.000 656 εργαζόμενους. Αυτό κύριοι Επίτροποι είναι το πρότυπο που απευθύνεται για τους εργαζόμενους στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Merci. Ε, ευχαριστώ. Pour la Commission économique et monétaire, Sven Sven τώρα από την Οικονομική και Νομισματική και μετά κάποιο μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης, κύριε Μόνασάκη. Ε, κύριος Γίγκολτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις σύντομες ερωτήσεις έχω μόνο. Πρώτον, η αξιολόγηση των συστάσεων αναχώρα ε, για το 2012. Δυστυχώς, οι δέσμοι που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δημοσίευσε μία εύληπτη επισκόπηση για το ποιες χώρες υιοθέτησαν τις περσινές συστάσεις και ποιες όχι. Γι' αυτό οι υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιφορτίστηκαν με αυτή τη δουλειά και σημείωσαν 140 συστάσεις περσινές, από τις οποίες μόλις 17 παρακαλώ ε, εφαρμόστηκαν πλήρως από τα μέλη του Συμβουλίου. Και θέλω να ρωτήσω, για ποιο λόγο δεν φτιάξατε ένα τέτοιο κείμενο, μια επισκόπηση ευανάγνωστη, εύληπτη και μπορείτε να μας πείτε, να δεσμευτείτε ότι θα το πράξετε έτσι ώστε να μπορούν τα μέλη του Συμβουλίου να βλέπουν πώς εφαρμόζουν τις, τις συστάσεις του. Δεύτερο, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει λέει μεταξύ άλλων στόχων και τους στόχους του προγράμματος για το 2020. Δυστυχώς τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο δεν αναφέρουν τους 7 στόχους κλειδιά και το τι έχουν κάνει τα κράτη, ε, ούτε το συσχετίζουν με το σχέδιο συστάσεων και πάλι οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκαναν αυτή τη δουλειά και είδαν ε, μεγάλες ανισορροπίες στις συστάσεις. 22 χώρες έχουν συστάσεις ε, για την απασχόληση, 9 για την καινοτομία, 8 για την ανεργία, και δύο μόλις για το περιβάλλον για τις εκπομπές διοξιδίου. Για ποιο λόγο αυτή η ανισορροπία και ιδιαίτερα οι επενδύσεις στο περιβάλλον γιατί δεν υποστηρίζονται περισσότερο παρόλο που είναι μια τεράστια ευκαιρία για την τόνωση ε, της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας. Και τέλος, πότε θα δημοσιεύσει την ανακοίνωσή της για την κοινωνική διάσταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό του Ιουνίου, γιατί έχω αυτή την περιέργεια. Ευχαριστώ. Ε, φαντάζομαι ότι είναι ερωτήσει που απευθύνεται και στου δύο επιτρόπους. Μάλιστα. Ναι. Η δεύτερη μάλλον προς τον κύριο Άντορ. Εγώ θα ήθελα να ακούσω την απάντηση και των δύο επιτρόπων, γι' αυτό ρωτάω. Η κυρία Μωρέν Σαρτιέ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Επίτροπη. Πρώτη ερώτηση με την ιδιότητα της μόνιμης εισηγήτριας για το ΕΚΤ αντελήφθην ότι έχετε κινητοποιηθεί βάσει των δηλώσεών σας τουλάχιστον για την ανεργία των νέων και από ό,τι κατάλαβα επικεντρώνεστε στις εγγυήσεις για τους νέους. Θέλω να επιμείνω σε ένα σημείο πρώτα απ' όλα. Σήμερα και ε, δοθέντως του αριθμού ανέργων νέων στο σύνολο της Ένωσης, παρότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες, ε, φρονείται πως είναι σκόπιμο να αυξήσετε το όριο ηλικία στα 30 χρόνια για τους ανέργους ε, νέους. Σήμερα είναι στα 25 χρόνια και ε, κατά αυτόν τον τρόπο ε, καλύπτεται το ίμιση των ανέργων. Εάν αυξήσετε το ηλικιακό όριο στα 30 χρόνια, συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μία ολόκληρη, ένας πολύ μεγάλος αριθμός νέων που δεν θα καλύπτεται από το νέο σύστημα Δεύτερον, ε, συνδυάζοντας την ανεργία με την οικονομική κρίση. Ε, ε, στον τομέα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ζητήσατε τις εγγυήσεις για τους νέους, την καταπολέμηση της φτώχειας, την απασχόληση για τους ηλικιωμένους, την απασχολησιμότητα του συνόλου των συμπολιτών μας με ποιο τρόπο μπορούμε σήμερα όλα να τα χώσουμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να βολέψουμε όλες αυτές τις πολιτικές. Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει στα ταμεία συνοχής ε, να ε, έχουμε ένα υψηλότερο κονδύλι για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το ποσοστό ε, του 25% δεν καλύπτει ε, τις τωρινές προτάσεις ε, για το 21-22%. Δεν είναι εφικτό. Ε, η κυρία Μπερές, πρωτού ακούσουμε τον Επίτροπο Αντόρ, θα ήθελα να καλωσορίσω την ομάδα προσκεκλημένων μου που εισήλθε στην αίθουσα, είναι από την προέρχονται από το ε, Ινστιτούτο Ζάκ Delors η Ευρώπη μας ε, και ασχολούνται με θέματα ε, ασφαλιών. Παρακαλώ κύριε Αντόρ, καλωσορίζω και εγώ τους προσκεκλημένους. Την Τετάρτη η Επιτροπή θα υιοθετήσει μια ανακοίνωση για την απασχόληση των νέων και θα έχετε έτσι πολύ περισσότερες προφορίες σε σχέση με αυτό που θα μπορούσα να σα δώσω σημερινή συνεδρίαση. Για να απαντήσω στην κυρία Μογάν Σαχτιέ, η διεύθυνση ανάμεσα στο ηλικιακό όριο 25 ή 30 έτη ε, και ε, φυσικά έχουμε και όλους όσους είναι πάνω από 25 χρονών και πρέπει να καλυφθούν από τα προγράμματα ε, πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούμε κατά προτεραιότητα με όσους είναι κάτω από 25 είναι ήδη πελώριο το έργο, χρειάζονται πολλές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο κρατών μελών και οι κρατικές υπηρεσίες απασχόλησης και όλοι όσοι εμπλέκονται στο σύστημα, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συνεργαστούν σε, με πολύ πιο εντατικού ρυθμούς. Εάν λειτουργήσει το σύστημα ε, εύρυθμα, τότε θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το ηλικιακό όριο. Το αρχικό μας σχέδιο που εγκρίθηκε από τους υπουργού και που περιγράψατε θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί για να ε, έχουμε κάποια απτή διαφορά σε κράτη-μέλη όπως η Γαλλία παραδείγματος χάρη ε, που ε, υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών εμπρος βάρος εκταμιεύουμε και στα πλαίσια πιλωτικών προγραμμάτων και νομίζω αυτό θα γίνει και στη δική σας χώρα. Ε, τώρα για την κοινωνική διάσταση. Δεν θα έρθει η ανακοίνωση αυτή την εβδομάδα. Εξαρτάται από τον πρόεδρό μας πότε θα το θέσει στην ε, ημερήσια διάταξη. Δεν μπορώ να προσθέσω κάτι άλλο σε σχέση με τις προηγούμενες απαντήσεις που έδωσα. Για το ε, ανελάχιστο μισθό στη Γερμανία και το δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung εκδόθηκε γερμανική δικαστική απόφαση και δεν την κατάλαβα τονίστηκε ότι όχι μόνο η έτσι Zeitung αλλά και άλλες εφημερίδες ασχολήθηκαν με το προηγούμενο και το τωρινό ευρωπαϊκό εξάμεινο και το πακέτο απασχόλης και τονίστηκε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ελάχιστο ε, μισθό για την ε, καταπολέμηση της ε, για τη βελτίωση της σχέσης με τη συνολική ζήτηση ε, και ε, υπάρχει μια ευρεία συμφωνία με την κυβέρνηση για αυτό το ζήτημα, όχι μόνο διότι είναι γενικώ αποδεκτό ότι οι μισθοί θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την παραγωγικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διότι είναι σημαντικό σε χώρες ουραγούς και όχι μόνο σε λίγα χρόνια, αλλά ε, με προοπτική μια δεκαετή περίοδο να παρέμβουμε, ώστε να διορθώσουμε ανισορροπίες Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλάβουμε αυτές τις πρωτοβουλίες για τη συνολική ζήτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, όχι μόνο για τις συγκεκριμένες χώρες. Ο πρόεδρος Μπαρόσο το ίδιο σημειωτώνησε κατά την παρουσίαση των ειδικών συστάσεων στα τέλη Μαΐου. Για τους περιβαλλοντικούς στόχους μιλήσατε για κάποια ανεπάρκεια Θα προσπαθήσουμε στο μέτρο του δυνατού στην προπαρασκευαστική περίοδο να καλύψουμε ε, κατά προτεραιότητα αυτή την ομάδα και σε συνεργασία με τον κύριο Ποτόσκι για θέματα περιβάλλοντος και αηφορίας και πράσινων θέσεων απασχόλησης να εξετάσουμε το τι θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε ε, στην υφιστάμενη διαδικασία. Ε, διαπιστώθηκαν όμως ανεπάρκειες και στον επόμενο κύκλο προγραμμάτων θα δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε την πράσινη απασχόληση ένα άλλο σχέδιο δράσης που ήταν στο πακέτο απασχόλησης για τις ε, θέσεις, ε, για τις νέες τεχνολογίες, έχει ήδη δρομολογηθεί ένας μεγάλος, ευρύς μάλλον, συνασπισμός. Και αυτό νομίζω θα συνεχίσει στην επόμενη ε, θήτια. Ευχαριστώ, Επίτροπος Ρεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Concerning, Mr. Ο Επίτροπος ε, Λάσλο Αντόρ ε, έδωσε ε, εξηγήσει για την ερώτηση που μου αφαιρούσε και εμένα. Εγώ δεν σχολιάζω τα σχόλια άλλων για τις ειδικέ συστάσεις για τη Γερμανία. Ε, συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με ημερομηνία 29 Μαΐου και αυτό θα λειτουργήσει ως βάση για τις μελλοντικέ εργασίες ε, της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Πρόκειται ε, για συμπεράσματα του Συμβουλίου. Για τον κύριο Τούσα, αναφέρθηκε στην τωρινή ε, κατάσταση στην ΕΡΤ. Στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου έδωσα μία απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν επεδίωξε το κλείσιμο της ΕΡΤ. Αυτό ε, θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών εξυγχρονισμού της οικονομίας της κυβέρνησης. Ε, αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη κατάσταση των εργαζομένων της ΕΡΤ και οι απολύσεις ε, ε, είμαστε σίγουροι ε, θα συνάδουν με το εφαρμοστέο νομικό ε, πλαίσιο. Εμείς υποστηρίζουμε την κρατική ραδιοτηλεόραση, θεωρούμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, παρότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να υποδείξεις της κυβερνήσεις το πώς θα πράξουν στον τομέα της ε, ραδιοτηλεόρασης. Ε, παρόλα αυτά τονίζει πόσο σημαντική είναι η δημόσια ραδιοτηλεόραση για την ελευθερία των ε, ΜΜΕ, την ποιότητα των ΜΜΕ, την πολυφωνία τους και τις δημοκρατικές αξίες. Ταχύτατα πρέπει να βρεθεί μια λύση το τελευταίο που χρειάζεται η Ελλάδα για κατοπέτραση η Ευρώπη είναι μια νέα κρίση. Κύριε Γκίγκολντ, τρεις ερωτήσεις θέσατε. Πρώτα απ' όλα, ποσοτικοποίηση της εφαρμογής των ειδικών ανάχώρα συστάσεων. Ε, πικροτούμε τις εργασίες του Κοινοβουλίου και της Γραμματείας της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ως προς την ποσοτικοποίηση της εφαρμογής. Πλην όμως είναι δυσχερές το έργο και θέλω να το τονίσω. Οι δημοσιονομικές πολιτικές ε, σχετικά εύκολα ποσοτικοποιούνται χρησιμοποιούμε δεδομένα από τη Eurostat και ε, οικονομικές προβλέψεις. Ταυτόχρονα για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αγοράς εργασίας, παραδείγματος χάρη της αγοράς προϊόντων, είναι στοιχεία ε, μάλλον ποιοτικά παρά ε, ποσοτικά. Δύσκολα λοιπόν μπορούν να να αναλυθούν από πλευράς ε, ποσοστών για να δοθούν συμβουλές σε όσους ε, εκπονούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, αλλά και τις εθνικές πολιτικές. Επιθυμούμε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αναβαθμίσουμε την μεθοδολογία ανάλυσης και τον τρόπο εκπόνησης πολιτικών. Δεύτερον, μιλήσατε για τις ανισορροπίες που διαπιστώνονται στις συστάσεις και αναφερθήκατε στις συστάσεις για το περιβάλλον και τις επενδύσεις. Η δράση και οι επενδύσεις στον τομέα του περιβάλλοντος έχουν ιδιαίτερη σημασία βράχει μακροπρόθεσμα διότι ε, τονώνουν την ανάπτυξη και επιτρέπουν την επιστροφή στην ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Σήμερα ήμουν στην πλατφόρμα για την αποτελεσματική χρήση των πόρων ε, και η πλατφόρμα αυτή τάχιστα θα εγκρίνει ένα έγγραφο συστάσεων για να βελτιώσουμε τις οικονομικές πολιτικές μας αξιοποιώντας καλύτερα τους υφιστάμενους πόρους μας. Είναι μια βραχυπρόθεσμη πολύ σημαντική πρόκληση στον τομέα αυτό. Τρίτη ερώτηση. Η κοινωνική διάσταση απάντησε ο Λάσλο Άντορίδη. Ήδη συνεργαζόμαστε για αυτό το θέμα και ε, θεωρώ ότι σύντομα θα καταλήξουμε και σε μια ανακοίνωση για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πάμε στο τέταρτο γύρο ερωτήσεων. Ξεκινάμε ε, από την ΕΚΟΝ, μετά από την, ο κύριος Σαματιάς και μετά η κυρία, ε, ο κύριος Σέρκας. Η κυρία Μαρίσα Ματίας, ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, να πω ότι μου φαίνεται ότι είναι ε, προφανές ότι εμείς ε, τη στιγμή που εγκρίνουμε ειδικέ συστάσεις θα πρέπει να κάνουμε και έναν απολογισμό των προηγούμενων στάσεων και του αντικτύπου τους. Και από αυτή την πλευρά μπορώ να θέσω δύο ερωτήματα. Πρώτον, εκπληρώθηκαν ναι ή όχι οι απαιτήσει των προηγουμένων συστάσεων από τις χώρες και δεύτερον, τα προβλεπόμενα αποτελέσματα επιτέχθησαν ναι ναι ή όχι. Ε, υπάρχουν διάφορα παραδείγματα για... Ε, αλλά ας πάρουμε την Πορτογαλία για το πρώτο ερώτημα. Εκπληρώθηκαν ή όχι οι συστάσεις. Γνωρίζουμε ότι οι ειδικέ συστάσεις ε, έχουν σχέση με την Τρόικα και το Μνημόνιο. Έγιναν 7 ε, διαδοχικές αξιολογήσεις και υπήρξε πλήρη συμμόρφωση. Σε σχέση τώρα με τα αποτελέσματα, τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, αν επιτεύχθηκαν ή όχι, εδώ διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα. Η ίδια η Τρόικα λέει το εξή. σε σχέση με το ΑΕΠ, ε, θα έχουμε ε, μείον 9 δις ε, για την ανεργία έχουμε διαφορά 5 ποσοστιαίων μονάδων και συνεχίζει με τα αποτελέσματα τι βλέπουμε ότι έγιναν αυτές οι προβλέψεις, οι οποίες ήταν εντελώς πλημελείς. Εάν λοιπόν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγνώρισε τα λάθη που έγιναν, ερωτώ τους επιτρόπους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αναγνωρίζει ναι ή όχι. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνει αυτή, ακολουθεί αυτή την οικονομική πολιτική ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γιατί κρίνει ότι οι νέε συστάσεις ε, θα οδηγήσουν στα αποτελέσματα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ διαψεύδεται στους ισχυρισμούς της από τα προηγούμενα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε Αλεχάνδρο Σέρκας και στη συνέχεια για την Επιτροπή. Ε, Κόνη, κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπη. Θέλω να δώσω την ε, ευκαιρία στον κύριο Ρε, να συνεχίσει να μας απαντά. Ό,τι και να γίνει κάθε χρόνο τις ίδιες συστάσεις φέρνεται. Αλλάζει ο ρυθμός, καλό είναι αυτό, ε, το τέμπο, αλλά η παρτιτούρα παραμένει η ίδια. Δηλαδή, και άλλη λιτότητα, και άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και άλλη εξυγίανση. Χιονίσει Χιονίση-βρέξη, ε, δεν παράνε κρίση ζήτηση, δεν παράνε κρίση χρηματοδότηση των μικρομεσών επιχειρήσεων. Και άλλες περικοπές και άλλη λιτότητα και μία από τα ίδια. Αλλά για μένα το σημαντικό ποιο είναι. Ό,τι και να γίνει στην πραγματικότητα, εσείς το χαβά σας. Αλλάζει ο ρυθμός, η μουσική όχι. Ποιος τη γράφει, ο συνθέτης ποιος είναι. Οι υπηρεσίες μας λέτε. Και τα γραφεία. Κοιτάτε και τα κράτη-μέλη καθόλου, φαντάζομαι. Βορείος του Ρήνου λίγο, έτσι, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλλά πολύ απλή ερώτηση. Το κοινοβούλιο τα ακούτε μια φορά ή μάλλον γιατί δεν το ακούτε το κοινοβούλιο ή τους πολίτες σε πάση περιπτώσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αδημοκρατικό σχέδιο. Μα ποιο εκπροσωπεί καλύτερα του πολίτε από το κοινοβούλιο μα. Το κοινοβούλιο σα είπε σταματήστε τι ασυμμετρίε και τι αποκλήσει στα κράτη-μέλη. Και ε, εσεί όλο και μεγαλύτερες αποκλήσει εισάγετε και τεράστια ρήξη μεταξύ του βορρά, του κέντρου και τη περιφέρεια. Και τώρα λέτε για τι συντάξει για την ε, ηλικία συνταξιοδότησης κάθε φορά και στη δική μου χώρα τώρα λέτε που είναι στα 67 να αυξήσουν και άλλο την ηλικία συνταξιοδότησης. Το Κοινοβούλιο μίλησε για ένα παράγοντα ε, ε, αηφορίας αλλά και ισότητας και δικαιοσύνης με τις συντάξεις. Αλλιώς θα γίνουν μεταρρυθμίσεις, λιτότητες, αλλά η ασφάλεια για πότε θα έρθει ε, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και συνδικάτα μας τα έχουν πει στο Κοινοβούλιο. Κύριε Ρεν, ποιον ακούτε ή γιατί δεν ακούτε το Κοινοβούλιο ή γιατί ακούτε πάντα τους ίδιους, εν πάση περίπτωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ και μετά η κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Πολύ σωστά δώσατε μεγάλη έμφαση σε σοβαρές διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάκαμψη και περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Ορισμένοι συνάδελφοι μίλησαν για το Βουνουτού στις παρεμβάσεις τους. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε τις διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις και την περικοπή των δαπανών. Ε, εξάλλου αυτά τα λέει και το Δουνουτού. Κύριε Σέρκας, θέλω να σας πω ότι και στην ε, Ελλάδα το όριο συνταξιοδότηση ε, είναι 67. Έτσι λέει η κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ε, στη Γαλλία όμως είναι 60. Υπάρχουν τεράστια χάσματα μεταξύ των χωρών. Το ερώτημά μου όμως είναι άλλο. Για τρία χρόνια τώρα έχουμε τις ειδικέ αναχώρασει στάσεις. Δύο χρόνια, εδώ και δύο χρόνια εφαρμόζουμε το six pack και πρώτη φορά, για πρώτη φορά εφαρμόζουμε το two pack. Όταν εξαρτάσετε ορισμένε χώρε, Φερρυπίν, Ολλανδία και Γαλλία, ε, παράταση της προθεσμίας για τους ε, δημοσιονομικούς στόχους. Αλλά οι συστάσεις για τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις είναι πάρα πολύ φιλόδοξες. Και για τη Γαλλία οι συστάσεις είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, πάρα πολύ ακριβείς. Πώς θα χρησιμοποιήσετε ε, τα εργαλεία που έχετε στο 2-pack και στο 6-pack για να ενθαρρύνετε την εφαρμογή των μέτρων. Το φθινόπορο, από ό,τι ξέρω, θα αναθεωρήσετε τα σχέδια προπολογισμών. Θα κοιτάξετε μόνο τα νούμερα, θα κοιτάξετε την ποιότητα επίσης των μέτρων που θα δρομολογηθούν. Τι, τι να περιμένουμε από εσά τους επόμενους μήνες και χρόνια. Ευχαριστώ. Ρετζίνα Μπάστος. Και μετά η Άννη Ποδηματά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω, μία προς τον Επίτροπο Ρεν και μία προς τον Επίτροπο Λάσλο Άντορε. Στην Πορτογαλία έγινε μία πελώρια προσπάθεια στον τομέα ε, των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών, ε, αλλά είναι εξαιρετικά αρνητικά τα αποτελέσματα. Ε, συμφωνώ ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει διευκολύνει την πρόσβαση στην πίστη, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι πρόσβαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το κόστος πιέζει την ευρωπαϊκή οικονομία και ιδιαίτερα την Πορτογαλία. Πέρα από τα μέτρα που αποφασίστηκαν στα πλαίσια του μνημονίου με την Τρόικα, ποια υπό άλλα μέτρα προτείνεται για την Πορτογαλία συγκεκριμένα. Επίτροπε Άντορ, στην Πορτογαλία ξέρετε ότι έχουμε από τα μεγαλύτερα ποσοστά ενεργεία των νέων στην Ευρώπη και ε, έχουμε ε, τώρα την προοπτική της των εγγύσεων των νέων. Ε, έχουμε άλλους μηχανισμούς ε, στη διάθεσή μας για την εγκατάλειψη του σχολείου από τους μαθητές και άλλες δράσεις στα πλαίσια του οικονομικού πακέτου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει άλλες απαντήσεις σε σχέση με όλους αυτούς τους μηχανισμούς ή θα περιοριστεί σε αυτές τις δράσεις. Σας ευχαριστούμε. Αν υποδηματά δύο λεπτά. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε της ε, Επιτροπής, θέλω να επανέλθω στο ερώτημα της εξαίρεσης από αυτή τη διαδικασία των συστάσεων ε, αναχώρα των χωρών που εφαρμόζουν πρόγραμμα σταθεροποίησης, τέσσερις το αριθμό σήμερα, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Κύπρος. Σας είχαμε πει πριν από καιρό μαζί με την συνάδελφο Φερέιρα ότι αυτή η εξαίρεση δημιουργεί προβλήματα προβλήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης και προβλήματα αποτελεσματικότητας γιατί δεν επιτρέπει μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων στο ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αλληλεπιδράσεις, τις επιτυχίες αλλά και τις αστοχίες αυτών των προγραμμάτων και για ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις. Σας είχαμε πει ότι αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα δημοκρατίας και το έλλειμμα δημοκρατίας δεν ευνοεί τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, την υπονομεύει και επειδή αναφερθήκατε στο θέμα της ΕΡΤ και επαναλάβατε αυτά που μας είπατε και στην Ολομέλεια, ότι δηλαδή επρόκειτο για μια αυτόνομη απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, να σας διορθώσω καταρχήν μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, όχι όλης της κυβέρνησης, γιατί η κυβέρνηση είναι τρικομματική, δεν είναι μονοκομματική. Και επίσης είπατε ότι στηρίζετε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στην Ελλάδα. Θέλω λοιπόν, επειδή αυτό επιδέχεται πολλών ερμηνεών, να σας ρωτήσω, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίζει αποφάσεις που παραβιάζουν βασικούς κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας χάρη της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος. Πιστεύετε ότι αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, ενισχύει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια ή την υπονομεύει. Και τέλος, επειδή επαναλάβατε ότι δίνεται σημασία στην ίση μεταχείριση όλων των κρατών μελών, Θέλω να σας ρωτήσω για άλλη μια φορά γιατί αρνείστε να εντάξετε τις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα στη διαδικασία των συστάσεων αναχώρα ώστε να υπάρξει ένας δημοκρατικός διάλογος για τα προγράμματα προσαρμογής και με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτές τις χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ. Θα αρχίσουμε αντίστροφα τώρα να απαντήσει πρώτο ο Επίτροπος ο κ. Ρέν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα αρχίσω ε, πρώτα από την ερώτηση της κυρίας Ματίας σε ό,τι αφορά την Πορτογαλία στην οποία και αναφερθήκατε. Η Πορτογαλία είναι χώρα σε πρόγραμμα όπως και η Ελλάδα και η Ιρλανδία. Έχει άλλη μεταχείριση. Ε, είναι τριμηνιές οι ε, επισκοπήσεις. Γι' αυτό διευκολύνει ε, τη ε, διαρκή αξιολόγηση του προγράμματος και των στόχων όσο και τη βελτίωση κάθε φορά του προγράμματος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του. Οπότε ε, αυτές οι τριμηνιές αναθεωρήσεις έχουν διπλό στόχο. Την παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος και στη συνέχεια το learning by doing. Δηλαδή, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία μας, προχωρούμε κάθε φορά. Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις αναχώρα είναι διαφορετικές. Η κυρία Ποδηματά αναφέρθηκε σε αυτό. Είναι αυτές οι τρεις χώρες. Οι χώρες που είναι σε προγράμματα θα πρέπει να συμμετέχουν στη γενικότερη διαδικασία των συστάσεων ε, στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και στο συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε πιστεύω. Ναι, όντως μπορούμε. Από την άλλη, δεν θα έλεγα ότι είναι μικρότερη η λογοδοσία. Έχουμε συνεχείς συζητήσεις και εδώ στην Επιτροπή σας και έχω απαντήσει ε, επί σειρά ετών πολύ συχνά στις ερωτήσεις σας και σε τακτά χρονικά διαστήματα για τις οικονομικές πολιτικές και ε, τα ε, προγράμματα οικονομικής προσαρμογής για τις χώρες που είναι σε προγράμματα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω το εξή και μάλιστα συνδέεται και με τον προηγούμενο γύρο ερωτήσεων και αυτό που ρώτησε ο κύριος Γκίγκολτ. συστάσεις για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας. Και η ιεράρχηση προτεραιοτήτων των προκλήσεων μπορεί να είναι συγκρίσιμη, αλλά όχι πάντα, γιατί ε, συχνά διαφέρουν οι πραγματικότητες από χώρα σε χώρα. Και δεν υπάρχει συχνά άμεση δυνατότητα σύγκρισης όλων των κρατών μελών στις περισσότερες περιπτώσεις. Αυτό δείχνει και μια αλλαγή στην προσέγγιση στο ευρωπαϊκό εξάμεινο σε σύγκριση με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Ο κύριος Σέρκας αναφέρθηκε στο ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει σχετική πρωτοβουλία πολύ σημαντική, διοργανώνοντας τις κοινοβουλευτικές ομάδες συνεδριάσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ε, και είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουν τα εθνικά κοινοβούλια περισσότερο και νωρίτερα σε εθνικό επίπεδο πριν εγκρίθει το εκάστοτε εθνικό πλαίσιο σταθερότητας και σύγκληση. Αυτό θα το καλωσόριζε πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή ίδια είναι πρόθυμη να κάνει συστάσεις χώρα και να συμμετέχει σε συζητήσεις με τα εθνικά κοινοβούλια για το σκοπό αυτό. Παρόλο που εδώ πρέπει να υπογραμμίσω ότι κατά κύριο λόγο αυτό είναι αρμοδιότητα του κάστο κράτου μέλου. Η κυρία Βόλτμαν Κόλ αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι συστάσεις θα παρακολουθούνται, θα ε, εξετάζεται η υλοποίησή τους. Απάντησα προηγουμένως στον κύριο Γκίγολτ σε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό το ερχόμενο φθινόπωρο να το συνδέσουμε και με την, ε, τον κανονισμό του Τούπακ για την ε, ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης και τους προϋπολογισμούς. Έτσι θα μπορούμε να ελέγχουμε καλύτερα ε, την υλοποίηση αυτών των συστάσεων και στη δημοσιονομική πολιτική αλλά και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αναφέρατε. Η απάντηση λοιπόν είναι καταφατική. Ε, το φθινόπωρο θα ε, αναθεωρήσουμε ακριβώς αυτές τις ε, συστάσεις και τον έλεγχό τους και θα τεθεί σε ισχύ και το 2 όπως είπαμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι θα μπορούμε να εκτιμούμε καλύτερα τους κρατικούς προπολογισμούς μετά τα μέσα Οκτωβρίου και είναι δικαίωμά μας όσο και ευθύνη μας να αξιολογούμε και τις δημοσιονομικές πολιτικές αλλά και τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις το πρώτο είναι πιο ποσοτικό, ένα το δεύτερο πιο ποιοτικό συχνά. Αλλά είναι σημαντικό να τα εξτάζουμε στο ίδιο πλαίσιο και να αναθεωρούμε και ε, να επισκοπούμε την ε, υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ε, είναι βραχυπρόθεσμες συζητάσεις και αφορούν ένα με τρία εξάμηνα. 6 με 18 μήνες. Αυτή τη στιγμή εγκριθούν από το Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ, ο κύριος Άντορ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είπε και ο κύριος Σόλι Ρεν, είναι πολύ σημαντικές για μας. Οι, εθνικ... Οι εθνικές απόψεις των Εθνικών Κοινοβουλίων επίσης είναι πολύ σημαντικές. Να σα δώσω, να σας το αποδείξω αυτό εμπειρικά. Συναντήθηκα με Γερμανούς ε, βουλευτές σήμερα από τη Τσεντεού. Πριν από λίγες εβδομάδες επισκέφτηκα το Λετωνικό Κοινοβούλιο και την επόμενη εβδομάδα θα είμαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στην Ελληνική Βουλή θα συναντηθώ με Έλληνες βουλευτές. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι συναντήσεις για να ανταλλάξουμε απόψεις για τις ειδικέ συστάσεις που αφορούν την εκάστοτε χώρα. Και δεν θα ξεχάσω και το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. Γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικές αυτές οι απόψεις. Μας το να συζητήσουμε μαζί τους την ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης και να προετοιμάζω, αφού έχω ακούσει τις απόψεις τους, ε, να προετοιμάσω τις ε, συστάσεις ε, και αφού έχω συναντηθεί με συνδικάτα. Επομένως πιστεύω ότι η δουλειά που κάνουμε βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις δημοκρατικές επαφές και ανταλλαγές απόψεων και θα συνεχιστεί αυτή η δημοκρατική διαβούλευση και θα ενισχυθεί αν γίνεται. Η κυρία Πάστας μίλησε για την Πορτογαλία. Την περασμένη εβδομάδα συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Πορτογαλίας στις Βρυξέλλες. Ο κύριος Μπαρόζο τον υποδέχτηκε και ήταν παρόντες και κάποιοι επίτροποι και όλοι και εγώ μάλιστα. Συζητήσαμε μάλιστα το θέμα της απασχόλησης και το θέμα της απασχόλησης κυρίως των νέων. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το συζητήσαμε. Αυτή τη στιγμή 90.000 νέοι θα υποστηριχθούν από αυτό το πρόγραμμα. Γίνονται και άλλες προσπάθειες για να αναβαθμίσουμε τη συμμετοχή της Πορτογαλίας στο σχήμα εγγύηση για την νεολαία. Ο κύριος Ρισάρα αύριο θα είναι στη Λισαβόνα και θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα. Ελπίζω λοιπόν όλες αυτές οι προετοιμασίες να οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα στο τελευταίο γύρο ερωτήσεων, η Οικονομική Επιτροπή καταρχήν, ο κύριος Φέιο, μετά η Άστριντ Λούλη και μετά από την Επιτροπή Απασχόλησης η Σιλβάνα Ράπτη και εγώ. Ο Διέγκο Φέιο πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να χαιρετήσω τους επιτρόπους Είμαστε σε ένα πολύ, σημαντικό σημείο των συζητήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωζώνη ειδικότερα. Γνωρίζουμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση ε, με την οικονομική ανάπτυξη, ε, με τη βελτίωση της κατάστασης στην αγορά εργασίας, κινήτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για την Ευρωζώνη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα ήθελα να γνωρίζω πώς, ε, ποια είναι η ανάλυση της κατάστασης ε, από πλευρά σας ε, των, χωρών που έχουν πρόγραμμα μνημόνιο. Ε, Παραδείγματο χάρη, η προσαρμογή για την ανεργία ήταν 12% και τώρα έχει φτάσει στο 18,5% με ποιο, πώς ακριβώς ερμηνεύεται τα αποτελέσματα αυτών των χωρών σε σχέση γενικότερα με την Ευρωζώνη και κυρίως εσείς κύριε Άντορο για την κατάσταση ως προς την ανεργία και τις βαθιές ανησυχίες που υπάρχουν σε αυτό τον τομέα. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω ποια είναι η θέση σας σε σχέση με τις δηλώσεις του κυρίου Ρασμούσεν ε, ο οποίος επέκρινε τις πολιτικές λιτότητας ε, σε σχέση με τους ε, προδιαγεγραμμένους στόχους. Στην περίπτωση της Ισπανίας, παραδείγματος χάρη, και αναφέρθηκε σε κλειδονισμού στην αγορά ομολόγων λόγω της πολιτικής λιτότητας. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το ζήτημα. Δεν πρέπει να μιλάμε με ένα, μία φωνή, δεν πρέπει να ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Ε, άρα εσείς πρεσβεύετε τις ίδιες απόψεις. Τι έχετε να πείτε. Η Άστριντ Λούλιν και η Σιλβάν Αράπτη ακολουθούν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Μία παρατήρηση γενική φύσεως θέλω να κάνω που αφορά τις αντιδράσεις των κυβερνήσεων στις ε, συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου μοιάζει οι κυβερνήσεις να αγνοούν τη διαδικασία. Διαδικασία που αποφάσισαν και οι ίδιες. Δηλαδή, ότι θα στέλνουν τα σχέδια προϋπολογισμού, τα προγραμματά τους, η Κομισιόν κάνει συστάσεις αφού τα αναλύσει και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικυρώνει. Αλλά ήδη τη στιγμή που η Κομισιόν δημοσιεύει αυτές τις συστάσεις, οι κυβερνήσεις κάνουν μούτρα, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, ε, για αυτά τα, τις επιταγές των Βρυξελών. Στη χώρα μου, ας πούμε, στο Μεγάλο Δουκάδο του Λουξεμβούργου, ο Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων είπε ότι με αυτές τις συστάσεις η Κομισιόν έχει χάσει το στόχο. Αυτός έχει χάσει τον μπούσουλα θα έλεγα εγώ. Εγώ θα ήθελα αυτές τις συστάσεις να είναι ακόμα πιο αυστηρές μάλιστα. Γιατί καλό θα ήταν για το μεγάλο δουκάτο να πούμε τα πράγματα ακόμα πιο ξεκάθαρα από ό,τι του τα λέμε. Και στη Γαλλία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανενδίαστα διαπίστωσε ότι δεν πρόκειται να σεβαστεί αυτές τις επιταγές. Αυτά είναι δημαγωγία. Σχιζοφρενία είναι. Σχιζοφρένεια, συγγνώμη. Στο Λουξεμβούργο ε, εξετάστηκαν αυτές οι στάσεις και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει τίποτα καινοφανέ σε σχέση με τις προηγούμενες. Και επομένω μια χαρά είμαστε εμείς στο Λουξεμβούργο, δεν υπάρχει λόγος να εκνευριζόμαστε. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να εκνευριστούμε και να διαπιστώσουμε ότι εφόσον υπάρχουν ίδιες συστάσεις σημαίνει ότι τίποτα δεν κάναμε εμείς ή δεν κάναμε αρκετά καλά τα πράγματα στο παρελθόν. Κύριε Αλούνη, σας παρακαλώ, όχι επιτρέψτε μου. Όχι, όχι, θέλω να δώσω το λόγο στη Σιλβάνα Ράπτη. Α, όχι, θέλω να αντιδράσουν, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχουμε τους οικονομικούς δείκτες, έχουμε τους οικονομικούς δείκτες για να βλέπουμε πώς πηγαίνει η πορεία με το έλλειμμα και το χρέος. Έχουμε τους κοινωνικού δείκτες για να βλέπουμε... Je peux continuer? Merci. Επαναλαμβάνω κύριε Ρεν, γιατί για σας κάνω την ερώτηση, δεν την κάνω για να ακούμε οι υπόλοιποι. Επαναλαμβάνω, έχουμε τους οικονομικούς δείκτες για να βλέπουμε πώς πηγαίνει η πορεία με το έλλειμμα και το χρέος. Έχουμε τους κοινωνικούς δείκτες για να βλέπουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις από τα προγράμματα λιτότητας τα οποία εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Ερωτώ, μήπως θα πρέπει να θεσπίσουμε και δίκτες δημοκρατίας για να βλέπουμε τι επίπτωση έχει στη δημοκρατία το κάθε πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος. Το ρωτώ αυτό κύριε Ρεν, γιατί ή κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε ή δεν καταλαβαίνετε πραγματικά. Ο Πρωθυπουργό Σαμαράς ξύπνησε ένα πρωί και χωρίς να ρωτήσει τη Βουλή χωρίς να ρωτήσει τους άλλους δύο εταίρους στην κυβέρνηση συνασπισμού, χωρίς να κάνει διαβούλευση με τους εργαζόμενους, καταπατώντας όλους τους κανόνες δημοκρατίας, έκανε ένα πραξικόπημα. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί σωστό, το αποδέχεται. Merci. Moi, je voudrais d'abord euh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ, κύριε Ρέν, καταρχάς να σας κάνω μια ερώτηση για τη σημασία που δίνεται στο λόγο των εμπειρογνωμόνων. Γιατί όταν σταματούν οι εμπειρογνώμονε να λέγουν αυτά που θέλετε εσεί να ακούσετε από τα χείλη του, θεωρείτε ότι δεν δικαιούνται δια να μιλούν. Παράδειγμα, ε, και τι εννοώ, το Δούνου του μπήκε στην Τρόικα διότι κάποια κράτη-μέλη θεώρησαν ότι ήταν ο καλύτερο τρόπο να ε, έχουν την καλή πραγματογνωμοσύνη και το καλό οδικό χάρτη για τις διαθωτικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και διορθώνει ε, τη γραμμή του, αναγνωρίζει τα λάθη του ε, στα μέτρα λιτότητας, πολλαπλασιαστές αλλά και ως προς το περιεχόμενο των διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων και ακούσαμε και τον κύριο Ρέγγιν και τον πρόεδρο Μπαρόζο να αποκηρύσει την νομιμότητα του Δουνουτού στην Τρόικα. Εσείς πώς το αξιολογείτε αυτόν τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζετε τους εμπειρογνώμονες. Εγώ είμαι από μια χώρα που έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη για τη δημοκρατία. Και κάθε φορά που οι διάφορες κυβερνήσεις, Ζουπέ, Σαρκοζή, προσπάθησαν να μεταρρυθμίσουν τις συντάξεις, το αποτέλεσμα ήταν πλήρης εμπλοκή τη κατάσταση στη χώρα και στου δρόμου, στι διαδηλώσει. Όπω γνωρίζετε, ο πρόεδρο Ολάντα από τότε που εξελέγει επανέφερε τον κοινωνικό διάλογο και ε, συζητούμε για το τι μέλη γενέστε και τι δεν γενέστε και στην αγορά εργασίας. Στις συστάσεις που κάνετε εσείς με τον κύριο Άντορ φρονείτε ότι προάγεται ο κοινωνικός διάλογος και ποια είναι η αντίληψή σας για την κοινωνική δημοκρατία. Ενώ ο κοινωνικός διάλογος είναι και ένα σημείο μάλιστα των συστάσεων ε, και των συμπερασμάτων ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τελευταίο θέμα. Είμαι έκπληκτη που δεν υπάρχει καμία σύσταση για τις ε, φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Ε, εάν θέλουμε μια στρατηγική για το 2020, μια φορολογία που ευνοεί τις κερδοσκοπικές κινήσεις και το βραχυπρόθεσμο κέρδος και να μην υπάρχει πουθενά σύσταση για τη φορολογία για τα κράτη-μέλη. Ε, να υπάρχει δηλαδή ένα φορολογικό σύστημα που να ευνοεί περισσότερο τις μακροπρόθεσμες ε, ε, επενδύσεις που τόσο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένω τις απαντήσεις σας, δεν ξέρω ποιος έλεξε κυρίες. start, immediately... Αν μου επιτρέψετε να απαντήσω και να αντιδράσω στο τελευταίο αυτό της φορολογίας που είπατε, από τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, την πατρίδα μου. Καμιά φορά ε, υπάρχουν δυσκολίες και αισθάνονται άβολα όταν μιλάμε για φορολογία. Και γίνονται αναφορές, ιδιαίτερα να φύγει η φορολόγηση από την εργασία ε, και, και προς τη χώρα που εσείς γνωρίζετε καλύτερα, τη δική σας πατρίδα έχουν απευθυνθεί τέτοιες συστάσεις, διότι είναι πολύ σημαντικό αυτό ε, σε καιρούς κρίσεων ιδιαίτερα για να τονωθεί η ζήτηση ε, για να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αυτό είναι σημαντικό ε, όταν υπάρχει ύφεση. Ε, στη συνέχεια, επανέρχομαι στην ερώτηση του κυρίου Φέιο που ρώτησε πώς ερμηνεύονται αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. 12% π.χ. ανεργία στην Ευρωζώνη, 11% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε, ε, αυτά είναι τα προβλήματα με το μέσο όρο. Ξέρουμε ότι είναι η ανεργία ρεκόρ, ο κόσμος το ξέρει, κατά μέσο όρο αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ουσία δεν φαίνεται από τα στοιχεία. Ποια είναι η ουσία, η πόλωση που υπάρχει πίσω από αυτό το μέσο όρο. Δηλαδή κάποια κράτη-μέλη ε, που είναι με στιβαρή οικονομία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, ε, με ανάπτυξη οικονομική την τελευταία διετία, ε, και ε, όπου αυξάνεται η απασχόληση. Από την άλλη έχουμε χώρες που έζησαν ε, τις επιπτώσεις κρίσης χρέους πολύ καιρό, παραμένουν σε ύφεση και άλλες και το χρόνου θα είναι σε ύφεση μάλιστα. Και εκεί η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται και μάλιστα η ανεργία των νέων ιδιαίτερα το τελευταίο έτος. Λοιπόν, εάν θέλουμε να βρούμε εδώ ένα αντίδοτο, δεν αρκεί να κοιτάμε τους μέσους όρους. Καλό είναι να έχουμε συστάσεις ε, ανά χώρα και ανομάδες χωρών. Γι' αυτό και στην παρουσίασή μας όλοι τονίσαμε την διαφορά ανάμεσα σε χώρες πλεονασματικές και χώρες ελληματικές, με διαφορετικά συμπεράσματα επίσης που πρέπει να εξαχθούν κάθε φορά από το διαφορετικό πλαίσιο. Αυτό επίσης κάνει να τονίζω ότι δεν ισχύει καθόλου ότι σε όλα τα κρατημέλη και στο σύνολο της Ένωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρεσβεύει ε, παντού λιτότητα και περικοπές. Σας είπα ότι πρόσφατα μετέβη στη Λετωνία. Η σύσταση εκεί είναι να διευρυνθεί κοινωνική ασφάλιση και βοήθεια. Ε, προηγουμένως μιλούσαμε για τη Γερμανία. Η σύσταση είναι πραγματικά εκεί να αυξήσουν τους μισθούς για διάφορους λόγους. Ε, κάνουμε λοιπόν ειδική ανάλυση ε, των καταστάσεων και των ε, ισχυουσών ε, συνθήκων σε κάθε χώρα. Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, και στο προηγούμενο κύκλο είχαμε τονίσει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανεργία των νέων. Αυτό ήταν πριν εγκριθεί η εγγύηση για την νεολαία. Τώρα έχουμε την εγγύηση για την νεολαία και πιο συγκεκριμένη εστίαση και δυνατότητα, όσο και υποχρέωση να δώσουμε αυτές τις συστάσεις στα ε, κράτη-μέλη για να μπορέσουν να εργαστούν για την εγγύηση για την νεολαία και όχι απλώς να αντιμετωπίζουν γενικά και αόριστα την ανεργία. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Διέγκο ε, Φέιου Εμείς υποστηρίζουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Το τόνισε αυτό. και το να διορθώσουμε το οικονομικό πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το θα υπάρξουν πολύ φιλόδοξοι στόχοι από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από τη Συνδοκορυφή, γιατί χρειαζόμαστε αυτή την όθηση για τη δουλειά που κάνουν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Εκομισιών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αναφερθήκατε στην κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προγράμματος. Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειε, θα ήθελα να τονίσω ότι μαζί με τις σχετικές κυβερνήσεις ετοιμάζουμε μία επιτυχή έξοδο από τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και για την Ιρτανδία και για την Πορτογαλία. Και στις δύο χώρες τα προγράμματα πάνε καλά και οι δύο χώρες επωφελήθηκαν πρόσφατα από τις αποφάσεις του Eurogroup σε ό,τι αφορά την παράταση της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων καθώς και τα επιτόκια. Εξετάσουμε και άλλες διευθετήσεις και προσαρμογές που μπορεί να χρειάζονται και να είναι χρήσιμες για να εξασφαλίσουμε ότι η έξοδος από τα προγράμματα θα είναι μια επιτυχής ιστορία και για την Ιρλανδία και για την Πορτογαλία. Αναφερθήκατε επίσης στις δηλώσεις του Γιώργ Γιάσμουσεν, ε, μέλος ε, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΑ. Δεν θέλω να σχολιάσω δηλώσεις μελών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μπορεί να το κάνουν τα ίδια τα άτομα αυτά. Ε, μπορείτε να δείτε το έγγραφο, το οποίο ε, είναι τμήμα του πακέτου που συζητάμε σήμερα. Η κυρία Άστριντ Λούλη αναφέρθηκε στις ε, ειδικές συστάσεις αναχώρα και τις συγκεκριμένες προς το Λουξεμβούργο, οι οποίες ήταν πολύ προσεκτικές και τις ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με μεγάλη σημασία, προσοχή και σημασία. Μιλήσατε για τις μεταρρυθμίσεις των συντάξεων. Είναι σημαντικό το Λουξεμβούργο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχουν τα δημόσια οικονομικά της ως προς τη βιωσιμότητά τους και εδώ ε, μπαίνει το πρόγραμμα των συντάξεων καθώς και των δαπανών γενικά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν μόλις το Δεκέμβριο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση και επομένως θα πρέπει το Λουξεμβούργο να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Παραδείγματο χάρη, τα μακροπρόθεσμα έξοδα θα συνεισφέρουν σε δύο ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το έξοδο, αυτά τα έξοδα, εν πάση περιπτώσει, ούτως ώστε ε, οι δαπάνες του Λουξεβούρου να είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο έχει προληπτικό χαρακτήρα. Εντοπίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και οι δράσεις που πρέπει να αναλυθούν πρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Ε, κοινωνικοί δείκτες. Σε αυτούς αναφέρθηκε η Σιλβάνα Ράπτη. Θα τους αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια της ανακοίνωσης για την κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Αναφερθήκατε στη δημοκρατία, που είναι μια βασική ευρωπαϊκή αξία. Και φυσικά εμείς ως θεματοφύλακες της συνθήκης φυσικά θέλουμε να υπερασπιστούμε αυτές τις θεμελιώδεις ε, δημοκρατικές αξίες. Η κρίση της Ελλάδας ήταν μάλλον αποτέλεσμα ανεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής και στατιστικών απατών. Πρώτα είχαμε την κρίση και μετά είχαμε το πρόγραμμα. Και η Κομισιόν μαζί με την ΕΚΤ και το Δούνου του, στα πλαίσια της πολιτικής εντολής που δόθηκε από, την το Ευρωγκρουπ Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα για την Ελλάδα, ούτω ώστε να επανέλθει σε τροχιά ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει η Ελλάδα, είναι σημαντικό η Ελλάδα, να εφαρμόσει το πρόγραμμα, προκειμένου να εξασφαλίσει ξανά την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και να αποφύγει την περιττή πολιτική αναταραχή, όχι μόνο για το δικό τη το καλό, αλλά και για το καλό όλη Ευρώπη. Τέλος για τις μεταρρυθμίσεις των συντάξεων και τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Ε, ακούστηκαν ερωτήσεις από την Πρόεδρο. Ξέρετε ότι εμένα με ενδιαφέρει τα μάλλα ο κοινωνικός διάλογος και οι κοινωνικοί εταίροι είναι σημαντικοί για να διευκολύνουν την νομιμότητα των αποφάσεων που θα πρέπει να έχουν πλατιά βάση. Η Γαλλία πάντα ήταν ε, πρωταθλητής του κοινωνικού διαλόγου. Αν και ορισμένοι το αμφισβητούν αυτό. Η Γαλλία πρόσφατα προοδεύει και συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου. Πιστεύω ότι μια πιστική μεταρρύθμιση των συντάξεων μπορεί να ετοιμαστεί χάρη σε αυτή τη μέθοδο με τη συμμετοχή δηλαδή, των κοινωνικών εταίρων. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι δεν δίνετε έμφαση στην αφορολογική μεταρρύθμιση. Ίσως ε, διαβάζουμε διαφορετικά έγγραφα. Εγώ έχω όμω τέτοιε συστάσει για διάφορα κρατημέλη για φορολογική μεταρρύθμιση, αν όχι για όλα τα κρατημέλη. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Για την ε, χώρα που ξέρω πολύ καλά μετά τη δική μου. Το Βέλγιο. Η σύστασή μα, η παριθμό 5, λέει για τη φορολογική μεταρρύθμιση. Γιατί το φορολογικό σύστημα εδώ στι Βρυξέλλε βασίζεται δυσανάλογα σε άμεσους φόρους. Και μπορούμε να αμφισβητήσουμε τη το κατά πόσο είναι δίκαιο αυτό το σύστημα. Το Βέλγιο έκανε κάποιε προσπάθειε να μειώσει το φορολογικό άχθο που βαραίνει τους εργαζόμενους, αλλά παρόλα αυτά ε, η φορολογία που βαραίνει τους εργαζόμενους ε, για τις περισσότερες θέσεις απασχόλησης, ε, περισσότερα είδη εργασία εν πάση περιπτώσει, είναι δυσανάλογα μεγάλο. Επίση υπάρχει πολύ ψηλή φορολογική, περιβαλλοντική φορολογία, συγγνώμη μπορούμε να απλουστεύσουμε κάλλιστα το φορολογικό σύστημα στο Βέλιο, να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά του, να απλουστεύσουμε τις φορολογικές δαπάνες, ούτω ώστε να συνεισφέρει και αυτό στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να εξασφαλίσουμε και μια κοινωνική δικαιοσύνη. Κυρία Πρόεδρε, Προσβλέπω στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με εσά, ούτω ώστε να προωθήσουμε αυτέ τι στάσεις για τη φορολογική μεταρρύθμιση και για τη μεταρρύθμιση των συντάξεων. Για να έχουμε και βιώσιμα δημόσια οικονομικά, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και για να αποκαταστήσουμε τα θεμέλια της βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ε, Ευρώπη. Ολοκληρώνεται εδώ αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να κάνω μόνο τα εξή δύο σχόλια. Πρώτον, ανεξαρτήτως της σημερινής ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα επ' ευκαιρία της παρουσίας των δύο επιτρόπων να σας πω πόσο αναστατωθήκαμε από αυτά που είπε ο κύριος Μπαρόσο ότι όποιος υποστηρίζει λέει, τη λεγόμενη πολιτιστική εξαίρεση είναι αντιδραστικός. Αυτό βλάπτει και μάλιστα με τρόπο υβριστικό το ευρωπαϊκό ιδεώδες και δεν αρκεί ε, ε, ένας εκπρόσωπος ε, να απαντήσει, θα πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Μπαρόσο. Ε, ε, οι δύο επιτροπές μας θα συνεχίσουν ε, την προσπάθεια και με τις δύο εισηγήτριες. Στις 9 Ιουλίου θα δούμε την έκθεση Φοντανέ, αλλά να σας πω τι νόημα έχει αυτό το εγχείρημα που κάνουμε εδώ, οι συστάσεις. Όλοι ανησυχούν για την ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου, για την ποιότητα αλλά και τη φύση της δημοκρατικής συζήτησης του διαλόγου. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα αν δεν εγγράφεται σε ένα πλαίσιο δημοκρατικό όπου ο καθένας να θεωρεί τον εαυτό του εταίρο και συμμετέχοντα της προσπάθειας που απαιτείται και της αλληλεγγύης επίσης. Πλην όμως, όταν εγκρίνετε εσείς αυτές τις ειδικέ συστάσεις αναχώρα, δεν ξέρω εκείνη τη μέρα τι ακριβώς άλλες υποχρεώσεις είχατε. Εγώ δεν βλέπω καμιά άλλη προτεραιότητα από το να έρθετε ακριβώς εκείνη τη μέρα που αποφασίζετε και δημοσιεύονται ε, αυτές τις συστάσεις αναχώρα να έρθετε να τις παρουσιάζετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λειτουργούν οι δημοκρατίες. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Αλλά ειλικρινά θα περίμενα και θα θεωρούσα ότι πέρα από τα λόγια η πραγματικότητα της δημοκρατικής λειτουργίας θα απαιτούσε άλλη οργάνωση και χρονική. Και ελπίζω του χρόνου, ανεξαρτήτως των διαφόρων ε, προβλημάτων που θα έχουμε λόγω των εκλογών ε, χρονικά και τα διάφορα ε, ημερολογιακά σκάμπα ανεβάσματα, θα μπορέσουμε ε, να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Σας ευχαριστώ και εξ ονόματος της Sharon Bowles και των δύο επιτροπών και κηρύσω το πέρα στη συνεδρία. ευχαριστώ.